Okay, we're going to open this meeting. Ας κηρύξουμε την έναρξη της συνεδρίας αυτής. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο Πρόεδρος! second. Witam Państwa i chciałem bardzo prosić za spóźnienie. Ja jestem pięć lat przewodniczącym tej komisji. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καθυστέρησα πρώτη φορά τα πέντε χρόνια τόσο πολύ. Δεν θυμάμαι στη ζωή μου να έχω καθυστερήσει τόσο πολύ, λέει αυτό μας στιγωνόμενος ο πρόεδρο. Εγώ φταίω. Πήγα στην Ιταλία σε αποστολή και μετά καθυστέρησε το αεροπλάνο και ε, τέτοια. Ερχόταν από τη Φραγκφούρτη, δεν προσγειωνόταν, δεν έφυγε στην ώρα του. Και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ για τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Είναι και η τελευταία συνεδρίαση. Λοιπόν, σε αυτή τη θητεία λάβαμε 6.000 αναφορές. Ε, κάθε χρόνο είχαμε περισσότερες αναφορές. Η Γραμματεία έλαβε περισσότερες από 12.000 επιστολές από διάφορους ετούντες. Ετοιμάσαμε 15.000 επιστολές εμείς, από τις οποίες οι 12.700 υπογράφτηκαν από μένα τον ίδιο. Ετοιμάσαμε πολλές εκθέσεις για την Ολομέλεια. Κάναμε πολλές αποστολές στην Ισπανία, στη Γαλλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, στη Μάλτα και στην Πολωνία. Επίσης, συμμετείχαμε στην προσωρινή επιτροπή για το Equitable Life και ακόμα ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή, ακόμα την παρακολουθούμε. Ο αριθμός των μελών πέρασε από τα 25 στα 40 σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο σέβεται το Κοινοβούλιο τη δουλειά μας. Εκατοντάδες ε, άτομα ήρθαν στις συνεδριάσεις ε, των επιτροπών, της Επιτροπής μας από όλα τα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά ε, συμμετέχαμε, συμμετείχαμε ενεργά για να βρούμε λύσεις για τις υποθέσεις. Είναι η μόνη κοινοβουλευτική επιτροπή που συνεργάζεται με τόσο απτό τρόπο με τους πολίτες της Ευρώπης. Θα ήθελα τώρα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, οι οποίοι συνεργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον διαμεσολαβητή και τους συναδέλφους τους και συνεργάτες του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που τόσο ενεργά δούλεψαν για να προωθήσουν τους στόχους της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι μετά από εμά ενδυναμώνεται αυτή η Επιτροπή, την αφήνουμε πιο ισχυρή, πιο καταξιωμένη και νομίζω ότι η επιτυχία της Επιτροπής μας οφείλεται και στη δουλειά που κάνει η Γραμματεία, ο Ντέιβιτ και η Κάρεν και οι συνεργάτες του, οι συνεργάτες τους που χωρίς αυτούς πραγματικά η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να είχε διακπαιριώσει όλο αυτόν τον όγκο δουλειά. Νομίζω ότι η αφοσίωσή του είναι το κλειδί τη επιτυχία μα. Του ευχαριστώ λοιπόν ολόψυχα. Θα ήθελα να πω επίση ότι οι προσπάθειέ μα να παραμείνουμε όσο τον πιο αντικειμενικοί στέφθηκαν από επιτυχία. Έτσι πιστεύω εγώ θα μπορούσα να παριθμώ επί ώρες τις υποθέσεις στις οποίες έχουμε εμπλακεί. Και συχνά βέβαια παίρναμε θέση υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, ε, κατανοούσαμε περισσότερο τον έναν από τον άλλο, αλλά τελικά παραμέναμε αντικειμενικοί. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μας επικρίνει κανείς για έλλειψη αντικειμενικότητας, για μεροληψία. Όχι, ήμασταν ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι. Θα συμφωνήσετε όλοι σας ότι δεν είμαστε ακριβώς ένα δικαστήριο, αλλά σχεδόν έτσι ένα παραδικαστικό όργανο και προσπαθούμε ως τέτοιο να είμαστε τόσο αντικειμενικοί όσο και οι δικαστές είναι ή θα έπρεπε να είναι. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι έχουμε επιτύχει σε αυτό το στόχο της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την ε, γραμματεία. Ούτε μία φορά αυτά τα πέντε χρόνια δεν μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η γραμματεία πρότεινε μία διαφορετική λύση από μια δίκαιη και τίμια λύση, προς την οποία κλείδαμε κι εμείς. Όλα τα μέλη της γραμματείας έδειξαν τρομερή εμπειρία και νομίζω ότι μοιράστηκαν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια σκιαγράφησης α, λύσεων. Σε αυτή, σε την προσπάθεια, συγγνώμη, της εξέβρεσης λύσεων. Και τους ευχαριστώ πραγματικά πολύ γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, και τώρα Πριν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για τη σημερινή μας συνεδρίαση, θα ήθελα να κλείσω διάφορες αναφορές. Μια πολο... πολωνικές αναφορές για την Βαλτική. Η έκβαση των αναφορών αυτών ήταν επιτυχής ε, για τους αναφέροντες. την 845, την 190 και όλες τις υπόλοιπες που έχετε στο έγγραφό σας. Αυτές θα πρέπει να κλείσουν, αυτές οι αναφορές, οι πολωνικές αναφορές επαναλαμβάνω. Επίσης μπορούμε να κλείσουμε τις εξή αναφορές από την Ιρλανδία. «908, 75, 160, 1673, και την ε, αναφορά για την προστασία του περιβάλλοντος στη Γερμανία. Έχουμε διάφορες αναφορές που θα συζητηθούν στο σημείο 7, 8 και 10. Παρουσία των αναφερόντων, καθώς και το σημείο 14. που επίσης είναι παρόντες οι αναφέροντες. Το σημείο 14 αφορά τους εκπροσώπους του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Κάποιοι όμως ε, Βούλγαροι βουλευτές δεν μπόρεσαν να έρθουν τελικά. Επίση, ε, θα συζητηθούν κάποια σημεία υπό το σημείο 19, αλλά όχι η παρουσία των αναφερόντων. Έχουμε μια άλλη αναφορά από την Πολωνία, μια άλλη αναφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσία των αναφερόντων. Τα σημεία 16 και 17 έχουν ακυρωθεί Επίση, όπω βλέπετε και στη μέση διάταξη. Με αυτέ τι αλλαγέ και τροποποιήσει, ελπίζω να συμφωνείτε να υιοθετήσετε την ημερήσια διάταξη ως προς την έγκριση της ημερήσιας διάταξης είναι νομίζω πολύ δυσάρεστο ότι στο τέλος θα έχουμε συντονιστές. Εγώ δεν μπορώ να παραστώ ούτε ο σοσιαλιστής συντονιστής και δεν είχε ανακοινωθεί εγκαίρως από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι θα γινόταν η συνεδρία των συντονιστών. Συγγνώμη σε Ρόμπερτ, αν μπορείτε να το ξαναπείτε, δεν είχα βάλει τα ακουστικά μου. Ναι. Μου φαίνεται αντιπαραγωγικό κύριε Πρόεδρε, πέμπτη βράδυ να κάνουμε συνεδρίαση των συντονιστών χωρί να έχει προηγουμένω ανακοινωθεί εγκαίρω. Εγώ δεν μπορώ να παραστώ και ο σοσιαλιστή συντονιστή επίση δεν μπορεί να παραστεί. Ξέρω ότι είναι φορτωμένη η μέρη σε διάταξη, αλλά αν δεν μπορέσω να θέσω τα θέματα που θέλω στους συντονιστές πρέπει να τα πω τώρα. Ίσως να μην είναι ο καλύτερος χρόνος, αλλά δεν βλέπω άλλη λύση. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω αφορά ένα αίτημα των κυρίων Ιταγκάη και Αγιάλα Σέντερ για την αναφορά 119208 όπου υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον μπορεί να είναι αποδεκτή. Δεν ξέρω τι φρονεί ακριβώς και η Επιτροπή και η Επιτροπή την απορρίπτει. Αυτό λοιπόν φρονούν και οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ και επομένως το θέτω. Το δεύτερο θέμα είναι ότι κάποτε πρέπει να συζητήσουμε τους διακανονισμούς, τις διευθετήσεις για το, την περίοδο από τώρα μέχρι την πρώτη την ιδρυτική μας συνεδρίαση. Τι θα γίνουν οι αιτήσει οι αναφορές που θα έχουν υποβληθεί εντωμεταξύ η γραμματεία μπορεί να μας εξηγήσει τι έχει προβλεφθεί ώστε να δούμε αν το δεχόμαστε. Για να απαντήσω στον Σερ Ρόμπερτ, όπως και τις προηγούμενες φορές που υπήρξαν ευρωεκλογέ. εφόσον συνεχίζεται η θητεία των παλαιών βουλευτών μέχρι τις 13 Ιουλίου, μέχρι ένα μήνα μετά τις εκλογές δηλαδή, θα πληροφορούνται τακτικά για σημαντικές αναφορές που έχουν υποβληθεί και η Γραμματεία θα διανύμει κατάλογο των αναφορών που θεωρεί ότι πρέπει να μπορούν να κλείσουν με τη θητεία αυτή, δηλαδή τις λεγόμενες αναφορές τύπου Β, που θα τις διανύμουμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και αν έχουν αντιρρήσεις να κλείσουν οι αναφορές αυτές με τη διαδικασία Β, αν έχουν αντιρρήσεις δεν θα κλείσουν και θα τις εξετάσει η επόμενη Επιτροπή Αναφορών μετά τις εκλογές. Αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει η εργασία μας απρόσκοπτα και να μην αντιμετωπίσουν οι καινούργιοι βολευτές έναν τεράστιο αριθμό καινούργιων αναφορών. Πρόεδρε, βεβαίως από τώρα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου ή οποτεδήποτε συσταθεί επισήμως η καινούργια Επιτροπή Αναφορών είναι πολύ στο καιρό. και εδώ μιλάμε για πέντε μήνες, έξι. Α, δύο δηλαδή. Α, καλά, ναι, αλλά για μένα οι δύο μήνες είναι σαν έξι. Λοιπόν, και από ό,τι κατάλαβα, εσείς μέχρι τη 13 Ιουλίου θα θεωρήσετε πρόεδρος. Μετά όμως θα υπάρξει δυσκολία, γιατί δεν θα επανέλθετε και μπορεί και άλλοι να μην επανέλθουν συνάδελφοι. Γι' αυτό θα ήθελα οι αναφέροντες να μην ζημιωθούν. Χαίρομαι που θα μας γνωστοποιήσουν ποιες αιτήσει θα έχουν υποβληθεί, αλλά μέχρι να συσταθεί επίσημα η καινούργια Επιτροπή Αναφορών και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι, δεν θα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Η Γραμματεία μόνο θα μπορεί να το κάνει και βέβαια είναι αντικειμενική διαδικασία για το κατά πόσο είναι αποδεκτή μια αναφορά ή όχι, αλλά αν υπάρχει κανένα κατεπήγον θέμα δεν μπορεί να αποφασίσει η γραμματεία. Τι θα γίνει τότε. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, κανονικά η θητεία διαρκεί μέχρι τις 13 Ιουλίου όπως είπα και πριν. Και αν όλα πάνε όπως έχουν προβλεφθεί τότε η θρητική της καινούργιας επιτροπής θα γίνει εκείνη την εβδομάδα. Μόνο μερικές εβδομάδες δεν θα υπάρχει επισήμως η Επιτροπή και το Προεδρείο της. Μερικές ημέρες λέω μόνο. Γιατί οι ιδρυτικοί και οι εκλογές, οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την εβδομάδα της 13ης Ιουλίου. Την πέμπτη το απόγευμα της ε, Συνόδου του Ιουλίου στο Στρασβούργο θα γίνουν ήδη αυτά. Άρα μόνο μερικές μέρες θα υπάρξει χάσμα. Κανονικά δε στην καινούργια θητεία την 1η και 2η Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής. Εάν όμως έχει προβλεφθεί, συμφωνούν οι καινούργιοι συντονιστές και ο καινούργιος πρόεδρος, μπορούν εκείνοι να συνεδριάσουν και μία εβδομάδα μετά την Ολομέλεια του Ιουλίου έτσι ακριβώς ώστε να δοθεί ε, κάποια πολιτική καθοδήγηση για το Σεπτέμβριο. Συγγνώμη πρόεδρε που επιμένω, αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε. Λέτε η συντακτική ε, συνεδρίαση να γίνει ε, την Πέμπτη το απόγευμα, αλλά ε, αυτό είναι στη φύση, στην πράξη αδύνατον, γιατί Όλοι θα έχουν φύγει. Εκτός από τους Γάλλου και τους Γερμανούς, οι φεύγουν. Οι πάντες φεύγουν. Έπειτα, θα υπά... αν γίνει συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα, δεν είναι κοινοβουλευτική ε, εβδομάδα αυτή. Μιλάμε για τις 28 Ιουλίου. Οι περισσότεροι θα έχουν πάει σε ακτές ή θα είναι σε διακοπές. Μέχρι τις 13 Ιουλίου δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί εσείς πρόεδρε θα είστε υπεύθυνο. Μετά τις 13 Ιουλίου, ο νέος πρόεδρος θα είναι εκείνος υπεύθυνο για την επίβλεψη και εποπτεία των αναφορών. Έτσι, δώστε μου την διασφάλιση αυτή. Αν ναι, αν έχω δίκιο, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Πρόεδρος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παρατείνουμε αυτή τη συζήτηση κυρίες και κύριοι, γιατί όλοι θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, μπορούμε να βρούμε μια λύση. Στην επόμενη συνάντησή μας. Μπορούμε να δούμε πότε θα κάνουμε αυτές τις αρχικές συνεδριάσεις, αυτές τις συντακτικές συνεδριάσεις, πότε θα οργανώσουμε τις επόμενες συνεδριάσεις. Ίσως η γραμματεία θα μπορούσε να μας στείλει και ένα email για αυτές τις δυνατότητε που έχουμε. Γιατί έχουμε εδώ διάφορου, διάφορους αναφέροντες ε, στην αίθουσα. Είναι κρίμα να καθυστερούμε τις ε, εργασίες μας, τις ουσιαστικές εργασίες μας. Η γραμματεία ας βρει τη λύση και ας στείλει ένα email σε όλους μας. Εντάξει. Concerning the, the question you raised about... Γραμματεία. Για την 1192 κάθετος 08 όλες οι ομάδες μετά από συνεννόηση μεταξύ τους συμφώνησαν ότι δεν είναι παραδεκτή αυτή η αναφορά. Πολύ ωραία τότε κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε και με τα διάφορα. Έτσι, με το σημείο 3. Έχουμε τον κώδικα ορθής πρακτικής που υπέβαλαν το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Αυτό το έγγραφο δεν διοθετήθηκε στην ε, τελευταία μας συνεδρίαση, γιατί ήταν πολύ λίγοι βουλευτές παρόντες. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και αν συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες, θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε τώρα. Εκτός και αν κάποιος θέλει το λόγο για αυτό το σημείο. Ο κύριος ο Σερ Ρόμπερτ, πρόεδρε. Δεν θέλω να παρατείνω αυτές τις συζητήσεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αναφέροντες εδώ που θέλουν να μιλήσουν. Γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά θα θυμάστε ότι αναβάλαμε αυτή τη συζήτηση την τελευταία συνεδρίαση γιατί ήταν πολύ λίγοι οι παρόντες. Ε, οι σοσιαλιστές που ήταν παρόντες ε, καταλαβαίνουμε ότι τότε δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν την άποψή τους. Τώρα όμως ε, μπορώ να πω σαφώς ότι οι σοσιαλιστές μέσω των συντονιστών δεν μπορούν να είναι παρόντες. Το συζήτησα με τη σοσιαλιστική ομάδα, μου επιβεβαίωσε ότι θα είναι κανένα εδώ. Οι δύο μεγάλες ομάδες, το ΕΛ και οι σοσιαλιστές, επιθυμούν αυτός ο κώδικας ορθής πρακτικής να γίνει αποδεκτός. Θα θυμάστε ότι υποβλήθηκε πριν από δύο ή τρεις συνεδριάσεις. Αμέσως μετά τις συζητήσεις που είχαμε την επόμενη μέρα σχεδόν. Δεν θέλαμε να αποκλείσουμε τις άλλες ομάδες, αντίθετα θέλαμε να συμμετάσχουν και οι άλλες ομάδες. Αυτό το κάναμε με στόχο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η Επιτροπή Αναφορών, με περισσότερους βουλευτές, με περισσότερους αναφέροντες παρόντες κτλ. Ο Αλεσάνδρο και εγώ και το προσωπικό μας, η βοηθή μας, δουλέψαμε πολύ σκληρά για να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι ευρέως αποδεκτό. Φυσικά, όταν διαδόθηκε στην αρχή, η εντύπωση που είχα είναι ότι τα υπόλοιπα μέλη ε, της Επιτροπής ε, γενικά μας υποστήριζαν και ότι δεν υπήρχε καμία διαφωνία, κανένα πρόβλημα με τον κώδικα ορθής πρακτικής. Λοιπόν, αυτά, αυτά έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, θα μπορούσα να επανέλθω αν υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν νομίζω. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν και άλλοι δύο βουλευτές. Και η κυρία Σίνοτ ζητάει το λόγο, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα δεν με έχει ικανοποιήσει η πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι δεν είναι σωστές οι διαδικασίες που προβλέψαμε. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει η έκθεση ονέστα που αντιφάσκει σε πολλά από αυτά που προτείναμε και από ό,τι έμαθα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και άλλων ομάδων στον καθορισμό της διαδικασίας ενώ εγώ απλώς έλαβα ένα κείμενο και δεν μου δόθηκε καμία ευκαιρία να το τροποποιήσω. Νομίζω λοιπόν ότι είναι λανθασμένη η ίδια η διαδικασία και η ομάδα μου δεν τη δέχεται. Όποτε θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά περιορίζομαι στα διαδικαστικά. Ε. Δεν ξέρω εσείς ως πρόεδρος τι λέτε. Ο κύριος ε, Χάμερστάιν στα αγγλικά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν ότι υπάρχουν στοιχεία και στις εκθέσεις Ονεστά και στην έκθεση Corbett που θα πρέπει να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια και που θα θέσουν ενδεχομένως, γιατί τα λέω αγγλικά, ε, ισπανικά πρέπει να μιλάω. Συγγνώμη, γυρνάω στα ισπανικά, το τσιπάκι δεν άλλαξα κάρτα σύμ. Λοιπόν, ε, μπαίνοντα τώρα στην ουσία του προβλήματος, βλέπω ότι υπάρχουν, λέω, και στην έκθεση Ονεστά και στην έκθεση ε, Κόρμπετ ε, προτάσεις για να βάλουν την Επιτροπή μας, να τις βάλουν ζουρλομανδία. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα για το Solvit και αλλού, θα το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλες προτάσεις τελείως αντιφατικές. Σε ό,τι αφορά τις διερευνητικές αποστολές εξεταστικές των πραγμάτων, επιτροπές για τις αναφορές σε άλλες χώρες, υπάρχει ο κανόνας, ο κώδικος συμπεριφοράς, ότι είναι μόνο περιγραφικές και τίποτα άλλο, δεν θα κάνουμε συστάσεις. Δεν υπάρχει πολιτικό ε, περιεχόμενο όμως εάν κάνουμε απλή περιγραφή της κατάστασης. Πολιτική επιτροπή είμαστε. Όταν κάνουμε τέτοιες αποστολές και επισκέψεις θα πρέπει να κάνουμε συστάσεις και ε, πληροφορίες. Δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ. Μου φαίνεται τελείως ε, ε, παρανοϊκή αυτή η πρόταση. Και θα πρέπει λέει, να έχουμε και εδώ συζητήσεις αντιφατικές με την πρόταση ονεστά που θα ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε το παραδεκτό ή μια ε, αναφοράς. Και άλλο φίλτρο λοιπόν θα βάλουμε σε αυτή την επιτροπή. Εδώ δεν μα φτάνει ο χρόνο να συζητήσουμε τι αναφορέ. Τώρα θα πρέπει όλε ολόκληρε να συζητούμε άλλα πράγματα, ε, εάν θα πρέπει να αποφασίσουμε όχι. Αυτό είναι ε, έλλειψη εμπιστοσύνη προ τη γραμματεία μα και του υπαλλήλου που πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσα να συνεχίσω κι άλλο επί τη ουσίας. Εγώ θέλω αυτή η συζήτηση να γίνει οπωσδήποτε την άλλη θητεία και να ξαναδούμε ακόμα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Σύνοτ, πολύ σύντομα. Αν κάτι είναι, λειτουργεί καλά, γιατί να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Μπορούμε όντως να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ανάγκες των αναφερόντων, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά πριν κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Σε Ρόμπερτ, να απαντήσω. Με ενοχλούν λίγο αυτά που λέει η κυρία Χάρκιν, γιατί αν θυμάμαι καλά, όταν η σοσιαλιστική ομάδα και το ΕΛΚΑ συνέταξαν αυτή την έκθεση. Ήταν ένα έγγραφο εργασία αυτή η έκθεση, στην πραγματικότητα. Το γράψαμε μέσα σε μία βραδιά και το υποβάλαμε την επόμενη μέρα στην Επιτροπή Προσυζήτηση. Δεν είχαμε σκοπό να αποκλείσουμε κανένα, έτσι. Αυτό το λέω ειλικρινά. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να αποκλείσουμε κανέναν. Το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές είναι η πλειοψηφία βέβαια. Αν είχαμε περάσει το θέμα στην Ολομέλεια θα είχαμε ήδη ξεμπερδέψει από τότε, αλλά δεν θέλαμε κάτι τέτοιο. Δεν θέλαμε να σας ε, εμποδίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, να σας αποκλείσουμε, αντίθετα. Αντίθετα, αν είχαμε πάει στην Ολομέλεια θα είχε περάσει το θέμα και θα είχε λήξει αυτή η ιστορία. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό. Με συγχωρείτε αλλά ζητώ να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Άτκινς προς τη γραμματεία και τους βουλευτές που έφυξε. Και εμείς ξέρουμε να διαβάζουμε, ξέρουμε τα κριτήρια και νομίζω λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη προς τη γραμματεία και τους συναδέλφους. Φτάνουν πια οι προσβολές εκ μέρους σας. Μα κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ Σιγά σιγά γίνονται ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Μην το ξεχνάτε. Και είναι μπροστά και οι αναφέροντες. Παρακαλώ να είναι όλοι ευγενείς και πεπολιτισμένοι. Μιλάμε για δεοντολογικό κώδικα εδώ πέρα, μια στιγμή, ο οποίος μπορεί να εγκριθεί μόνον αν συμφωνούν όλοι, αν τον δέχονται όλοι δεν είναι επίσημο έγγραφο που να απορρέει ε, άμεσα από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου ούτε είναι τίποτα το υποχρεωτικό το οποίο να πρέπει να εφαρμόσουμε ούτως ή άλλως. Μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαδικασία που προτείνεται, μπορούμε να την απορρίψουμε. Άρα βλέπω ότι οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ φαντάζομαι ότι δέχονται τη διαδικασία γιατί οι φιλελεύθεροι η πράσινη και η κυρία Σίνωτ ε, ενώ η πράσινη η φιλελεύθερη και η κυρία Σίνωτ είναι κατά άρα δεν μπορούμε να το δεχτούμε δεν μπορεί να εγκριθεί άρα το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να οργανωθεί μια άλλη συζήτηση για τη γραμματεία ή για τις διαδικασίες δεν μπορούμε όμως να χάσουμε άλλο χρόνο σήμερα για αυτό το θέμα δεν βλέπω καμία δυνατότητα έγκρισης τη διαδικασία τώρα, όση ώρα και να το συζητήσουμε. Κύριος Χα... Όχι, ο Σερ Ρόμπερτ. Μα εγώ μιλούσα κύριε Πρόεδρε και ζητήθηκε διαδικαστικό, με διέκοψαν δηλαδή. Συνεχίζω λοιπόν. Εγώ Πρόεδρε ποτέ δεν είπα τίποτε άλλο, όπως και οι σοσιαλιστές, δεν έκανα καμία αξιολογική κρίση, δεν είναι αμφιλεγόμενο θέμα και γι' αυτό με εκπλήσουν αυτά που είπαν οι δύο καλοί μου αυτοί φίλοι και συντονιστές των άλλων ομάδων. Το γεγονός παραμένει ότι η Γραμματεία διένει με αυτό το έγγραφο και από τη σύντομη συζήτηση της τελευταίας φοράς όπου δεν ήταν οι συνάδελφοι αυτοί παρόντες είχε γίνει προσπάθεια να φανεί ότι το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές προσπαθούν να στριμώξουν τους υπόλοιπους. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν συζητήθηκε ποτέ το έγγραφο αυτό. Το να λέτε λοιπόν ότι εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό είναι λάθος. Απλώς ποτέ δεν το συζητήσαμε. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό όμως. Και δεν δέχομαι τις κατηγορίες που ακούστηκαν. Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής μας είναι συλλογικός. Εάν ορισμένοι συνάδελφοι δεν δέχονται οτιδήποτε προτείνεται και δεν θέλω εδώ να σας ε, ανησυχήσω ή να μαλώσουμε Ούτε προσπαθώ να κοροϊδέψω κανέναν. Δεν είναι τέτοια η φήμη μου εξάλλου. Εδώ υπενήσονται ότι γίνεται ελιγμός και δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ξέρω ότι ο Ντέιβιντ δεν δέχεται αυτό που ακούσαμε, έχει είναι δικαίωμά του. Νομίζω πάντως κύριε Πρόεδρε ότι για να προχωρήσουμε θα πρέπει να αποσύρω το έγγραφο αυτό και ζητώ να συζητηθεί άλλη φορά. Δεν θέλω να τροποποιηθεί αλλά να επανυποβληθεί με τον δέοντα τρόπο όποιες ομάδες το εγκρίνουν και να συζητηθεί όπως πρέπει. Γιατί μέχρι τώρα δεν συζητήθηκε ποτέ πράγμα για το οποίο δεν ευθύνομαι εγώ. Μα δεν υπήρχε απαρτία την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει. Ωραία. Θα κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος ε, ο Σερ Ρόμπερτ όταν η νέα ε, επιτροπή συσταθεί, έτσι, στο νέο κοινοβούλιο. Σημείο 5. Έχουμε ένα έγγραφο για την επίσκεψη που έγινε στο Gateshead και στο Newcastle. Πρόκειται για την αφορά 727-2005. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να μιλήσει για αυτό το σημείο. Ναι, ο κύριος σήκωσε το χέρι του. Στα αριστερά μου. Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μιλήσει για αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθούμε την κατάσταση ε, για αυτή την χιτά. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα για τις υδρογεωλογικές συνθήκες της χιτά. Ε, η έκθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες Βρετανικές αρχές. Ε, ζητούν να έχουν το χρόνο για να γίνει μία ενδελεχής εξέταση. Είμαστε σε επαφή με τις Βρετανικές αρχές για να δούμε σε τι συμπέρασμα θα φτάσουν από αυτή την έκθεση για τις υδρογεωλογικές, υδρογεωλογική κατάσταση. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες από τις αγγλικές αρχές, ε, θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τη διαδικασία. Οι αναφέροντες ήταν πολύ, έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από την επίσκεψη της Επιτροπής και ελπίζουν ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή, ούτω ώστε οι κατάλληλε αρχές να δώσουν την απάντηση που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Φυσικά και δεν θα κλείσουμε την αναφορά αυτή. Μετά από αυτά που μας είπε η Επιτροπή, απλώς κλείνουμε μία φάση της διαδικασίας, δεν κλείνουμε όμως την αναφορά. Φαντάζομαι λοιπόν, θα συμφωνείτε με τα όσα λέει η έκθεση, πολύ ωραία, και μπορούμε να αφήσουμε αυτό το σημείο και να πάμε στο σημείο 6. Αναφορά 686 του 2006. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αναφέροντας είναι ο το μέλος του Συνδέσμου Εμπόρων και Εισαγωγέων Αυτοκινήτων της Ελλάδας Πρόκειται για ένα σύνδεσμο που καλύπτει διάφορες μάρκες αυτοκινήτου. Η αναφορά αυτή παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2006 και εν συνεχεία δόθηκαν και περαιτέρω ε, κείμενα στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο κάποιοι εισαγωγείς, επίσημοι εισαγωγείς έχουν ε, παραβιάσει τις αρχές ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Οι αναφέροντες παρουσίασαν στις 21 Δεκεμβρίου του 2006 ένα παράπονο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια αναφορά, με βάση το διαδικαστικό κανονισμό 1 του 2003, με τα ίδια επιχειρήματα που είχε και η αρχική αναφορά. Σε αυτό το παράπονο, αν θέλετε, σε αυτή την ε, δεύτερη αναφορά, μας ενημερώνουν ότι έχουν υποβάλει και αντίστοιχη αναφορά στις ελληνικές αρχές ανταγωνισμού. Η Κομισιόν για αυτό το παράπονο θεώρησε ότι ακόμη και αν οι πρακτικές αυτές αποδειχθούν, οι πρακτικές που καταγγέλει ο σύνδεσμος, δεν αφορούσαν παρά μόνο την ελληνική επικράτεια, το ελληνικό, τον ελληνικό χώρο. Αυτές οι πρακτικές δεν εντάσσονται σε ένα σύνολο, σε ένα πλαίσιο που θα έφυγε και άλλα κράτη-μέλη. Επομένως, οι πολιτικές και οι πρακτικές αυτές που καταγγέλλονται, ακόμη και αν αποδειχτούν, δεν θα συνιστούσαν κοινοτικό θέμα, κοινοτικό ενδιαφέρον, μια και οι επιπτώσεις θα αφορούσαν μόνο την ελληνική επικράτεια και καθόλου τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Επομένως, οι αρχές της Κομισιόν σημείωσαν ότι ο σύνδεσμος απλώς υπέβαλε ε, μία αναφορά σε εμά και βεβαίως και στην αντίστοιχη ελληνική αρχή ανταγωνισμού. Οι ελληνικές αρχές ανταγωνισμού λοιπόν ήρθαν σε επαφή μαζί μας και διαπιστώσαμε ότι η αναφορά που έλαβαν ε, οι ελληνικές αρχές κάλυπταν όλα τα στοιχεία της αναφοράς που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, οι δύο αναφορές είναι πανομοιότυπες. Η Κομισιόν ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές να ασχοληθούν αυτές με το θέμα αυτό. Απάντησαν ότι μπορούν να το κάνουν. Η Κομισιόν, ήρθαν ξανά, η Κομισιόν ήρθε ξανά σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και οι ελληνικές αρχές μας είπαν ότι ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Η Κομισιόν λοιπόν αποφάσισε να απορρίψει για αυτό το λόγο την αναφορά που της υπευλήθη. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν το Δεκέμβριο έγραψαν μια επιστολή προς τους αναφέροντες, Δεκέμβριο του 2007, εξηγώντα την κατάσταση. Είναι... Τους εξηγήσαμε δηλαδή ότι το θέμα αυτό είναι θέμα της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου δεν απάντησε σε αυτήν την επιστολή που στείλαμε του Δεκεμβρίου 2007 και επομένως στις 5 ε, Μαρτίου του 2008 η Κομισιόν απέρριψε την αναφορά του Συνδέσμου με βάση τον ε, κανονισμό, τον διαδικαστικό κανονισμό. Στο άρθρο αυτό, στο άρθρο 13, η Κομισιόν ε, μπορεί να απορρίψει μία αναφορά όταν ασχολείται με την αναφορά αυτή η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού. Επομένως έχουμε αρχιοθετήσει εμείς αυτή την ε, αναφορά και δεν σκοπεύουμε να ξανασχοληθούμε με την αναφορά αυτή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροφής. Αυτά Πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ματσούκα. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να προτείνω, επειδή έχουμε κάποια ζητήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εάν θα ήταν εφικτό να τα συζητήσουμε όλα μαζί για να μην επανερχόμαστε διαρκώς με την Επιτροπή. Θέλω μόνο επί της ε, συγκεκριμένης αναφοράς ε, να ρωτήσω την Επιτροπή με ποια ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συνομίλησε και συνεννοήθηκε. Διότι δυστυχώς η χώρα μου τα τελευταία χρόνια πλήττεται από πληθώρα σκανδάλων, μέσα σε αυτά και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προσωπικά δεν είμαι καθόλου περήφανη για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο θα ήθελα και με αφορμή τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της Επιτροπής να την καλέσω να δει πιο σοβαρά τις υποθέσεις αυτές, όπως επίσης να την καλέσω να δει πιο σοβαρά και το δικό της έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Εάν δεν παρεμβαίνει πιεστικά όπου βλέπετε ότι υπάρχει κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση ή καρτέλ, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αλλά και σοβαρές ευθύνες προς εσάς. Ευχαριστώ. Με ευχαριστώ. Μήπως θέλετε να απαντήσετε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση αυτή. Ε, Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων και καλείται να συνεχίσει αυτό το ρόλο της στα πλαίσια των όσων ορίζει η ε, κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δράση της. Αυτή η κείμενη νομοθεσία είναι κυρίως κανονισμός 1 του 2003 ο οποίος ορίζει ένα σύστημα καταμερισμού εργασίας σύμφωνα με το ε, κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού και είναι αρμόδιο από τη μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει για να επιβάλλει ανάληψη δράση σε μια αρχή ανταγωνισμού προκειμένου, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική αρχή ανταγωνισμού όντως, όντως ε, ακολουθούσε, ε, παρακολουθούσε εκ για την ε, υπόθεση αυτή. Και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κυρία Ματσούκα, σας ρώτησε κάτι πολύ συγκεκριμένο όμως. Ποια είναι αυτή η αρχή με την οποία εσείς συνομιλείτε στην Ελλάδα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό. Ναι, έχουμε αυτή την ενημέρωση. Είναι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, λένε στα αγγλικά οι Έλληνες ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ορίζει το άρθρο 35 του κανονισμού 1 του 2003. Και με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως πάντα, ήταν η επαφή μας. Πριν αρμόδια αρχή. Κυρία Ματσούκα, παρακαλώ. Ναι, αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η οποία βεβαίως επιμένει να υποστηρίζει και να διατείνεται ότι συνομιλεί με μια ανύπαρκτη και διαλυμένη και διεφθαρμένη Ελληνική Επιτροπή ε, κατά τούτο και επειδή είναι ένα μείζον ζήτημα, πιστέψτε με αντιλαμβάνομαι τη θέση στην οποία βρίσκεστε, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε κι εσείς τη θέση στην οποία βρίσκονται οι αναφέροντες. Ε, τα εργαλεία που διαθέτουμε είναι πάρα πολλά, οπότε θα προτείνω να τα αξιοποιήσουμε όλα. Πάντως για τη συγκεκριμένη αναφορά προτείνω να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρότεινα λοιπόν να αφήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή και υποθέτω και προσβλέπω στη συνέχιση της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο σημείο 7. Είναι η αναφορά υπέρ 130 του 2007. Παρευρίσκεται ο αναφερομένος κύριος Γεώργιος Φλωράς. Έχετε 5 λεπτά παρακαλώ. Στα αγγλικά, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου. Προτιμώ να το πω στα αγγλικά. Θα αρχίσω παραθέτοντας τρεις γραμμές από το Your Europe που είναι στο σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δίκαιος ανταγωνισμός είναι ε, κεντρικός για την πολιτική της Ένωσης και την ανάπτυξη. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει όρους για δίκαιο και ανοιχτό ανταγωνισμό στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια ε, για ε, τη διασφάλιση του θεμητού ανταγωνισμού χωρίς τρευλώσεις και διορθώνει ε, αντίστροφες συμπεριφορές. Στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται όλα αυτά. Βάσει της δαμοθεσίας αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι Εφτά χρόνια κάθε περίπτωση κάνει να ολοκληρωθεί και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονό ότι είναι μεγάλη περίπλοκη ελληνική αγορά. Η επίσημη δικαιολογία που δίνει η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι έχουν έλλειψη προσωπικού. Και ρωτούμε, ποιο αποφασίζει για τη στελέχωση, για την πρόσληψη νέου προσωπικού στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού οι ε, ολιγορίες ε, νομίζουμε εμείς ότι είναι εσκεμμένες, χρονοτριβούν και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού ε, δείχνουν προκλητική αδιαφορία να στελεχώσουν την επιτροπή αυτή για να μπορεί γρήγορα να αντιδρά και να δρά. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ορίζει ότι κάθε εθνική αρχή ανταγωνισμού πρέπει να είναι εξάρτητη. Αυτό τι σημαίνει. Ότι θα πρέπει να έχουν την εξουδότηση να κάνουν τι απαραίτητε ενέργειε έτσι ώστε να λειτουργούν γρήγορα και σωστά. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού μόνο ανεξάρτητη δεν είναι και υποστελεχώνεται διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αποφασίζει να του αφήσει να κάνουν τι απαραίτητε προσλήψει. Παρόλο που είναι μεγάλη πρικοδότηση δεν προσλαμβάνουν προσωπικό. Για το λόγο αυτό και ως αποτέλεσμα έχουν τεράστιες καθυστερήσεις στο έργο του. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει γενικό διευθυντή από το Σεπτέμβριο του 2006. Δυόμιση χρόνια χωρίς γενικό διευθυντή. Και ισχυρίζονται ακόμα ότι κάνουν αυτό που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Δυόμιση χρόνια χωρίς γενικό διευθυντή. Κεφάλαια έχουν όμως για να αγοράζουν γραφεία που κοστίζουν 14 εκατομμύρια ευρώ. Το ευκαταφρόνητο αυτό ποσό. Σήμερα εκτός από τη δική μου εταιρεία έχουν έρθει και άλλοι Έλληνες πολίτες εδώ που έχουν προσφύγει κατά πολυεθνικών γιγάντων όπως είναι η Fiat και η Nestlé. Η εταιρεία μου στράφηκε κατά της Oxford University Press και της Pearson που είναι ε, μεγάλοι εκδότες, γίγαντες εκδότες. Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορούμε να περιμένουμε 7 χρόνια απέναντι σε αυτούς τους γίγαντες. Είναι παράλογα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια τέτοια καθυστέρηση τι σημαίνει ότι όποιο τολμάει να τα βάλει με τα καρτέλ θα τον σβήσουν από την αγορά. Αυτό είναι αντικίνητρο για όποιο προτίθεται να στραφεί κατά τον καρτέλ. Δεν είναι τυχαίο που τα καρτέλ κυβερνούν και διοικούν και βασιλεύουν στην ελληνική αγορά. Είναι η ε, ευρωπαϊκή χώρα με τις υψηλότερες τιμές σε σχέση με το εισόδημα των πολιτών. Η ε, Επιτροπή Ανταγωνισμού πάντα πατώνει στις διεθνείς αξιολογήσεις. Η δική μου εταιρεία πριν από τρία χρόνια είχε 75 εργαζομένους και σήμερα 45 μόλις. Από το 2001 στο 2006 καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσει μας κατά 300%. Σήμερα οι πωλήσει μας έχουν φτάσει σε επίπεδα του 2005. Μας ε, περιφρονούν ως επιχειρηματίες και ως ε, πρόσωπα. Από υπερήφανοι ε, επιχειρηματίες τώρα δανειζόμαστε από γνωστούς φίλους και προμηθευτές. Γιατί, γιατί δεν παίρνει απόφαση η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Η άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λέει ότι δεν μπορεί να υπαγορεύσει τα κράτη-μέλη πόσο χρόνο χρειάζεται για να ελέγξουν κάθε περίπτωση ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, κάποια κράτη-μέλη σαν την Ελλάδα δεν προσλαμβάνουν αρκετό προσωπικό, άρα ε, έχουν μεγάλε χρονοτριβέ και καθυστερήσει. Προτείνουμε να ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα στελεχώνεται κάθε Επιτροπή Ανταγωνισμού Εθνική, λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμό της κάθε χώρας και άλλα σημαντικά στοιχεία. Έτσι, κάθε χώρα δεν θα μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη δικαιολογία της υποστελέχωσης για να παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού. Απευθύνουμε έκκληση προς εμάς να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 226 επί παραλήψη εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού. Απευθύνουμε έκκληση σε εσά. Υποτίθεται η κυβέρνηση ότι εφαρμόζει τον νόμο. Θυμίζουμε ότι το 10 επανειλημμένα όρισε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την εσωτερική τους ένωμη τάξη ως δικαιολογία για τις καθυστερήσεις. Άρα και οι δικαιολογίες της ελληνικής κυβέρνησης ότι έχουν μεταφέρει την νομοθεσία δεν ευσταθούν, διότι δεν εφαρμόζεται. Είναι λογικό δηλαδή κατά την ελληνική κυβέρνηση να περιμένουμε και 20 και 30 χρόνια μέχρι να δεήσει να αποφασίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή τύχη στις επερχόμενες ευρωεκλογέ. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Χιώτη και την ομάδα της και το επιτελείο για τη βοήθειά της. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από άλλους αναφέροντες ή αναφερόμενους για άλλες αναφορές να μιλήσουν πρώτα και μετά να γίνει μια γενική συζήτηση και των τεσσάρων. Σερ Ρόμπερτ. Να κάνω μια ερώτηση. Λέει ο Σερ Ρόμπερτ, τι στο καλό είναι αυτή η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και τι κάνει, μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει, σας παρακαλώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω θα μπορούσε να μας εξηγήσει, απαντώντας μόνο σε αυτή την ερώτηση του Σερ Ρόμπερτ. Τι επιτροπή είναι αυτή, τι θεσμός είναι αυτή η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρακαλώ δώστε μας μια σύντομη απάντηση. Και όχι επί της ουσίας της αναφορά παρακαλώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1 του 2003 για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού υπάρχει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών. Οι Εθνικές Αρχές μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούν από κοινού αυτό που λέγεται δίκτυο ECN ένα δίκτυο το οποίο συνεργάζονται οι αρχές για να εφαρμόζεται το δίκαιο ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος οργανισμός είναι αυτός, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ε, είναι μια επιτροπή που απαρτίζεται κυρίως από δύο ταχύτητες, ή δύο επίπεδα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος προτείνει τις αποφάσεις ε, και μετά υπάρχει και έναν ε, δικαστικό σώμα που είναι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από τον Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σταύρος Σαρής έχει το λόγο. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ε, έχω κάνει την καταγγελία από το 1997. Χρειάστηκαν 12 ολόκληρα χρόνια για να βγει μια απόφαση, η οποία βγήκε πριν 16 μέρες. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρά τις οχλήσεις μου όλα αυτά τα 10 χρόνια, πότε τελικά θα αρχίσει να ερευνάτε, δεν έβρισε καμία ανταπόκριση. Αυτό συνέβη μόνο όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο τύπος άρχισαν να γράφουν για τις καθυστερημένες υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δυστυχώς όμως, ο ρόλος και η υποχρέωση οποιασδήποτε επιτροπής ανταγωνισμού είναι να επιλαμβάνεται άμεσα ή σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν κάποιος καταγγέλει πρακτικές και όχι να κάνει 12 χρόνια. Στην προηγουμένη περίπτωση στη δική μου τι έγινε. Έγινε μια νεκροψία. Όταν κάνω μια νεκροψία είναι μεταφορικό φυσικά αυτό το οποίο λέω, ή ο καταγγέλων έχει πεθάνει, ή η επιχείρησή του έχει καταστραφεί. Εγώ καταστράφηκα, η επιχείρησή μου. Εγώ ζω ακόμη. Η απόφαση η οποία βγήκε δεν με ικανοποιεί, διότι ενώ έχω καταγγείλει στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πρακτικές της ΦΙΑΤ οι οποίες είναι ίδιες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση απάλλαξε την εταιρεία Fiat SPA, την Ιταλική τη μητρική, όπως απείλαξε και την Fiat Credit. Θα ήθελα να αναφέρω έτσι να δείτε τι γινόταν όταν ζήτησα η, Επιτροπή, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με έγγραφό μου να με ενημερώσει την πορεία της. Το έγγραφο αυτό είναι 23 Τετάρτου του 7. Θα σας το δώσω μετά. Στο οποίο αναφέρεται όλα αυτά τα χρόνια τι γινόταν ο φάκελό μου. Μεταφερότανε από προϊστάμενο σε άλλον προϊστάμενο, από υπάλληλο σε άλλον υπάλληλο και ποτέ όμως κανένας δεν άνοιξε αυτή την καταγγελία και να κάνει την έρευνα. Και θα προτίμωσα πολύ και θα ήταν πολύ καλό να ασχολιόταν και να έλεγε η Επιτροπή ότι δεν έχει βάση η καταγγελία σας, μπαίνει αρχείο. Ποτέ δεν πήρα αυτή την απάντηση. Επειδή όμως η καταγγελία μου από το 1997 ήταν έγκυρη. Ήτανε για παραβάσεις ανταγωνισμού πρακτικών και πολιτικών της ΦΙΕΤ δικαιώθηκα μετά από 12 χρόνια. Το πρόστιμο το οποίο επευλήθη για μένα είναι ένα χάδι που κάνανε. 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Παραλείψανε πολλές παραβάσεις που έχω καταγγείλει και γι' αυτό μετά από 10 μέρες ετοιμάζω δεύτερη καταγγελία. Είχα στείλει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνισμού δύο επιστολές γιατί δεν επιλαμβάνεται, γιατί δεν στέλνει κάποιον εκπρόσωπο να δει τι γίνεται με την υπόθεσή μου. Σας έχουν απαντήσει οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στην αναφορά μου ότι μόνη αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή. Θέλω να θυμίσω όμως ότι έχω κάνει και μία προκαταγγελία τον τέλος Οκτωβρίου του 2008 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαταγγελία για πολιτικές και πρακτικές που γίνονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης πανομοιότυπε με την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στο σημείο 9. 103. Ο κύριος Λαφαζάνης, 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι ε, ε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, παρουσιάζουμε εδώ ενώπιόν σας ως εκπρόσωπος της εταιρείας Γεώργιος Δρίτσας που δραστηριοποιείται δεκαετίες τώρα στην Ελλάδα στο χώρο της επεξεργασίας και πώλησης καφέ. Είμαστε εδώ διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να σας μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας ώστε αυτές ενδεχομένως να ληφθούν από εσάς υπόψη για μια βελτίωση της λειτουργίας των κανονισμών ανταγωνισμού ανά την Ευρώπη. Η εταιρεία μας το 2002 κατήγγειλε την ΕΣΤΛΕΣ την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος για παραβάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού. Χρειάστηκαν 7 χρόνια μέχρι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βγάλει απόφαση. Συγκεκριμένα έβγαλε απόφαση το Φεβρουάριο του 2009 καταδικάζοντας την ΕΣΛΕ για παραβάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού και επιβάλλοντας ένα πρόσημο 30 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα 7 χρόνια η Επιτροπή Ανταγωνισμού παραβατικά ολιγορούσε και η Εστλέ σε όλο αυτό το διάστημα αλώνιζε την ελληνική αγορά εκμεταλλευόμενη τον Έλληνα καταναλωτή αλλά και καταπιέζοντας με κάθε τρόπο και οποιονδήποτε μικρότερο ή μεγαλύτερο ανταγωνιστή της και πετυχαίνοντας να ελέγχει το 93% της ελληνικής αγοράς του καφέ στην Ελλάδα. Ε, στο μεταξύ διάστημα και μέχρι να βγει η απόφαση δεχθήκαμε εκατοντάδες μηνύσεις και αγωγές από την Νεστλέ που στόχο είχαν την εξουθένωσή μας οικονομικά και ηθικά. Μετά ε, από αγωγή μας η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταδικάστηκε σε πρόστιμο για την ολιγορία της με 30.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι ε, συμβολικό αλλά δείχνει ότι η παραβατική συμπεριφορά της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναγνωρίστηκε και από ελληνικό δικαστήριο. Μηνύσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για παράφαση καθήκοντος και η εκδίκαση θα γίνει το 2010. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι όπως όλα δείχνουν ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά από το μεγάλο διεθνές κεφάλαιο και αυτό επιβάλλει τους όρους με τους οποίους η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί όπως επίσης επιβάλλει και τη στελέχωσή τη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ιδρύθηκε με κάποιο νόμο το 1977. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει 17 διαφοροποιήσεις πάνω σε αυτό το νόμο. Έως το 2007 η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είχε εκδώσει καμία απόφαση. Αποφάσεις άρχισαν να εκδίδονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της οποίος ήρθε από την Ευρώπη στην Ελλάδα και ο οποίος ξέθλαψε τις ξεχαμένες όλες υποθέσεις από τα συρτάρια με σκοπό να ε, ε, εξεταστούν αυτές τις υποθέσεις. Τέτοιες υποθέσεις είναι του κυρίου Σαρή, η δική μας και άλλες πολλές. Με το που άρχισαν να εφαρμόζονται όμως οι πρώτες καταδικές αποφάσεις ε, για παραβάσεις του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, άρχισαν και οι προσφυγές των καταδικαστέντων στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτά κατά τεκμήριο δεν γνωρίζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο οι αποφάσει τη Επιτροπή Ανταγωνισμού όλο και περισσότερο να αμφισβητούνται από τα διοικητικά εφετεία. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη αρχή και ποιο είναι το κύρος της. Εάν οι κανόνες του ανταγωνισμού κρίνονται ουσιαστικά στα διοικητικά εφετεία, τότε πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να είναι περιττή ή είναι αναγκαία για αυτούς οι οποίοι την ελέγχουν ώστε να με τη συμπεριφορά της και τις καθυστερήσεις της να οδηγεί σε ε, καθυστέρηση των τελεσίδικων αποφάσεων ώστε στο μεταξύ διάστημα και τα διαστήματα αυτά από ό,τι ακούτε είναι πολλών ετών η, τα μονοπόλια να λειτουργούν εις βάρος του καταναλωτή. Πίστη μας είναι ότι ιδιαίτερα σε μικρές και διαπλεκόμενες δυστυχώς... Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πάμε στο σημείο 10. Ο κύριος Κοσμόπουλος. Πέντε λεπτά όμως, παρακαλώ μην υπερβαίνετε το λεπτό σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριοι Ευρωβουλευτές που είχατε την... Ε, ε μας δίνετε μάλλον τη δυνατότητα να παρευρεθούμε σήμερα εδώ και να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Βρίσκομαι εδώ υπό δύο ιδιότητες. Εκπροσωπώ την εταιρεία Aerotenco, μια εταιρεία ε, λιανικής πώλησης σιδήρου στην Ελλάδα, αλλά συγχρόνως είμαι και με την ιδιότητα του Προέδρου της πρώτης και μοναδικής μέχρι στιγμής αντιμονοπολιακής οργάνωσης της Ευρώπης, της Ένωσης Θυμάτων Καρτέλ και Μονοπωλίων που είναι γνωστή με την επωνυμία Stop Cartel. Με αυτή λοιπόν τη διπλή ιδιότητα έρχομαι σήμερα πολύ φορτισμένος και πολύ θυμωμένος κύριοι σε αυτή την αίθουσα. Και είμαι φορτισμένος και θυμωμένος διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία κατέφερε το χωρίς προηγούμενο, ακριβώς κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τενέζος, Διευθύνων Σύμβουλος της καταγγέλουσας εταιρείας για την οποία σας μίλησα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 77η ημέρα απεργίας πείνας την οποία πραγματοποιεί έξω από το κτίριο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Αθήνα. Καταφέραμε δυστυχώς το ακατόρθωτο. Ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Τενέζος και θα παρακαλούσα το Σεβαστό Προεδρείο να μου δώσει λίγο χρόνο παραπάνω να μιλήσω για αυτό το συγκλονιστικό γεγονός το οποίο προσβάλλει τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Ο Ευρωπαίος αυτός πολίτης, ένας σας διαβεβαιώ αξιοπρεπέστατος μικρομεσαίος επιχειρηματίας, έφτασε στην εσχάτη αυτή μορφή διαμαρτυρίας ακριβώς για τους λόγους τους οποίους ακούσατε αυτή τη στιγμή από τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους μου που ήρθαμε σήμερα στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ σοβαρό κύριε Πρόεδρε και κύριοι Ευρωβουλευτές το γεγονός αυτό να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Είναι η συμπεριφορά την οποία επί 77 μέρες επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση επικέστατα χαρακτηρισμένη σαν προκλητική, βάρβαρη, απολύτιστη πολιτική συμπεριφορά. Και αυτή έχω έρθει σήμερα κατηγορηματικά και εν γνώση του τι λέω να καταγγείλω ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσω παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι η τελευταία θεσμικά δυνατότητα την οποία έχετε να συνεδριάζετε να εξαντλήσετε κάθε διαδικαστική δυνατότητα ούτως ώστε να καταδικαστεί αυτή τη στιγμή αυτό το πολιτικό φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης στην Αθήνα του πολιτισμού στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα του πολιτισμού και το οποίο αφήνεται να εξελίσσεται ανάγκητα από μια κυβέρνηση η οποία επί 77 ημέρες δεν έχει αρθρώσει μία λέξη κύριε. Πολύ σύντομα θα με συγχωρέσετε τόσο για την ένταση όσο και για το αίτημά μου να έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ το γιατί ο κύριος Στενέζος, ο Ευρωπαίος αυτός πολίτης, βρίσκεται επί 77 μέρες σε απεργία πείνας μπροστά στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο προμηθευτής του, η μεγαλύτερη χαλιβουργική εταιρεία της Ελλάδος, ευνηδίως, χωρίς να υπάρχει κανένας εμπορικός ή οικονομικός λόγος, του διακόπτει την προμήθεια το καταγγέλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού του ζητάει στοιχεία ρωτώντας τον εάν κατά τη δική του γνώση ως μέρος της αγοράς υπάρχει καρτέλ χάλιβα στην Ελλάδα. Προσκομίζει επισήμως τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δηλαδή προσκομίζει πίνακες ολόκληρους συνεχών από το 2000 και δόθε παραλίλων μεταβολών των τιμών πωλήσεως του χάλιβα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και από τις τρεις χαλιβουργίες προσκομίζει κουστούνια ολόκληρα ε, τιμολογίων που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό. Περιμένει λοιπόν μετά από δύο σχεδόν χρόνια κύριε πρόεδρε θα ήθελα να μου δώσετε ε, το να Proszę pana, jedna minuta, ale to Ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό αυστηρά, ένα λεπτό. Μιλάτε όλοι για το ίδιο θέμα. Κατανοώ πραγματικά βαθύτατα ε, το πρόβλημά σας, αλλά τα επιχειρήματα επαναλαμβάνονται. Ένα λεπτό σας, παρακαλώ πολύ. Το μικρόφωνο σας. Κοιτάνε πάνω. Η Επιτροπή λοιπόν Ανταγωνισμού στην Ελλάδα αντί να διερευνήσει το σύνολο της καταγγελίας βγάζει μία εισήγηση και μετέπειτα απόφαση η οποία ασχολείται με το 10% της καταγγελίας και αφήνει ανέπαφο την καταγγελία για την ύπαρξη και λειτουργία καρτέλ στην Ελλάδα. Υποβάλλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αντί αυτή να γίνει αντικείμενο εισήγησης και απόφασης της Ολομέλειας Επιτροπής Ανταγωνισμού απορρίπτεται προσωπικά με απόφαση προσωπική του Προέδρου. Αυτά και μόνον και πολύ συνοπτικά είναι τα αίτια διότι ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε στην απόγνωση έχοντας και πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως προείπαν και οι συνάδελφοι εδώ Κάθε άλλο παρά ανεξάρτητη είναι, διορίζεται στην ουσία από τους μεγαλοκεφαλαιούχους οι οποίοι ελέγχουν την ελληνική... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ε, ας το οργανώσουμε το εξ, ως εξής. Έχουμε εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, παρόντα, εδώ. Τα άκουσε όλα αυτά. Έχουμε και ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ίσως σύντομα να μιλήσει και μετά σύντομη συζήτηση. Παρακαλώ εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτές, ε, καλησπέρα σα. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Ονομάζομαι Γιώργος Καπανταϊδάκης. Ε, είμαι εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, υπεύθυνο για θέματα βιομηχανική πολιτική ομολογώ ότι συμμετέχω για πρώτη φορά σε παρόμοια συνεδρία, αντικαθιστώντα συνάδελφο ο οποίο απουσιάζει για υπηρεσιακό λόγο στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι παρακολούθησα με ενδιαφέρον ε, τις παρατηρήσεις των ε, αναφερόντων. Έχω καταγράψει λεπτομερώς τις παρατηρήσεις τους και τις μεταφέρω στο κέντρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα παρέμβω. για την αναφορά 96-2008 του κύριου Σαρή, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή τον Ιανουάριο του και μετά τον Μάρτιο του 2008. Και εμείς το απαντήσαμε σύντομα τον Απρίλιο. Του εξηγήσαμε ότι υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ημών και των εθνικών αρχών. Και με βάση αυτό το σύστημα καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, οι ελληνικές εθνικές αρχές είναι οι αρμόδιες για να παρέμβουν όταν αυτές οι συμφωνίες αποκλειστικής ε, εμπορικής διάθεσης έχουν επιπτώσεις ε, αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Επίσης, η Εθνική Αρχή μπορεί να αποφασίσει να βάλει τέλος ε, στις παραβιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ασχοληθήκαμε με την αναφορά του κυρίου Σαρή και κάναμε ένα καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Ελήφθησαν κάποια ασφαλιστικά μέτρα και τελικά το Μάρτιο του 2009 πήρε απόφαση η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως είπε και ο κύριος Σαρής. Θα ήθελα να σας πω ότι είπαμε τον Απρίλιο στον κύριο Σαρή, δηλαδή ότι, ότι αν η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει τη δουλειά της, ούτως πίν, και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα κράτη-μέλη, υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια δικαστική έρευνα. Αυτή η δικαστική έρευνα έγινε στην περίπτωση του κυρίου Σαρή. Μας ενημέρωσε ο κύριος Σαρής το Μάρτιο για αυτό το θέμα. Και του είπαμε ότι ένα ελληνικό δικαστήριο λοιπόν θα ασχοληθεί με τη συμπεριφορά της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού, που είναι η επιτροπή αυτή, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτά για την αναφορά 96 ε, 2008 του κ. Σαρή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε. Αν λένε όλοι ότι ο καθένας έκανε το καθήκον του, δεν μου επαρκεί αυτό σε εξήγηση. Κυρία Ματσούκα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ε, ειλικρινά λυπάμαι που σήμερα στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής αναφορών για αυτή τη θητεία ε, συζητάμε τόσο σοβαρά και σημαντικά ζητήματα. πιστέψτε με αυτές οι πέντε αναφορές που συζητώνται σήμερα είναι ένα ελάχιστο δείγμα για να αντιληφθείτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι πολλές περισσότερες οι περιπτώσεις, οι σχετικές περιπτώσεις με τις ε, αναφορές που συζητούμε σήμερα. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή του αναφέροντε και του καλωσορίζω, του συμπατριώτε μου σήμερα στι Βρυξέλλε. Θα ήθελα να του καλωσορίζω για έναν άλλο λόγο, πιο καλό και πιο θετικό, παρά για να ακυρώνουμε ουσιαστικά ε, την ευρωπαϊκότητα της Ελλάδας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκανε μια παρένθεση, μια παρέκκληση από τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια και σύντομα θα επανέλθει. Υπάρχουν και οι θεσμοί και η βούληση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ε, από τους αναφέροντες και κυρίως θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις στην, ε, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ανταγωνισμός, ε, κυρίες και κύριοι, αποτελεί το συστατικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς και η εσωτερική αγορά αποτελεί τον βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να έχουμε λοιπόν υγιή και ωφέλιμο ανταγωνισμό, και για όλους προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι και να τον παρακολουθούμε και να τον ρυθμίζουμε. Εδώ λοιπόν είναι ο ρόλος σας. Ο ρόλος σας θα πρέπει να γίνει πιο σκληρός ε, και σαφώς ε, η έλεγχη που θα κάνετε να είναι πιο ουσιαστική. Και μιας και είμαστε σε περίοδο ευρωεκλογών, να σας ε, μεταφέρω κάτι που συμβαίνει νομίζω στα περισσότερα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη υπάρχει ως άλοθη στους κυβερνώντες όταν κάτι δεν πάει καλά να λένε ότι φταίει η κακή Ευρώπη. Αποδείξτε λοιπόν εσείς πριν από όλους, που έχετε και την αρμοδιότητα, ε, ότι η Ευρώπη λειτουργεί σωστά, παρακολουθεί τους κανόνες, ρυθμίζει την αγορά και αποδίδει το δίκαιο σε όσους πολίτες αδικούνται στις χώρες μέλη. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για εσάς. Θα πρότεινα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, και κλείνω εδώ, αφού σας ευχαριστήσω για την ε, πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και εσάς και τη Γραμματεία και όλους τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα για τα συγκεκριμένα ζητήματα να ζητήσω να παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ, καθώ επίση, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σα ζητήσω να υπογράψετε τι ε, επιστολέ που θα στείλετε εσεί στι ελληνικέ αρχέ, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω και να απαντηθούν στην Επιτροπή Αναφορών οι συγκεκριμένε ε, υποθέσει. Σα ευχαριστώ θερμά. Πρόεδρε, μου φαίνεται ε, πραγματικά εξαιρετικό αυτό που σημαίνει έκτακτο και τρομερό. Πέντε αναφορές ακούσαμε και την ουσία συζητούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται ε, το θέμα ε, είναι στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση προηγουμένως σε αυτή την ε, επιτροπή έχουμε μεγάλη εμπειρία από τέτοιες υποθέσεις όπως με το Equitable Life όπου δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν ή να συνειδητοποιήσουν ότι υπήρχε πρόβλημα. Και όχι μόνο οι ρυθμιστικές αρχές δεν κατάλαβαν ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος όπως στην ε, Βρετανία και στην Ελλάδα αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Άκουσα λοιπόν αυτές τις παρεμβάσεις που ήταν έτσι πολύ έντονα φορτισμένε και δεν με εκπλήσει αυτό γιατί δημιουργήθηκαν τεράστιες ζημίες ε, λόγω της μεγάλης ανικανότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τα γεγονότα. Εμεί ω Επιτροπή Αναφορών δεν έχουμε την εξουσία του το δικαίωμα να παρέμβουμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι η δουλειά μα αυτή. Η δουλειά μα είναι να αντιδράσουμε ε, στα παράπονα που εκφράζουν ε, οι πέντε αυτοί διαφορετικοί άνθρωποι και να ε, ρωτήσουμε την Επιτροπή τι κάνει για αυτό το θέμα. Δεν έχω την εντύπωση και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η διακεκριμένη Αντιπρόεδρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει. Ε, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο και στο παρελθόν. Γι' αυτό, Πρόεδρε, σας κάνω έκκληση να κρατήσετε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να ενημερώσετε την Επιτροπή ή να την παροτρύνετε, αν θέλετε, να κοιτάξει πιο προσεκτικά το πώς λειτουργεί αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν κάνει τη δουλειά της. Και θα είναι λάθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι λάθος που έχει φτάσει ήδη στο επίπεδο που έχει φτάσει το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο λοιπόν. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Με, μετά από όλα αυτά που είπε ο Σερ Ρόμπερ και η κυρία Ματσούκα, θα γράψουμε μια πολύ αυστηρή ε, επιστολή στην ε, Επίτροπο κυρία Κρός, που είναι η αρμόδια Επιτροπή για τον Ανταγωνισμό και θα αφήσουμε όλες αυτές τις αναφορές ανοιχτές. Ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτό θα σας δώσω για όλους σας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα λεπτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω 4-5 σχόλια σύντομα. Η Κομισιόν δεν απεκδίεται των ευθυνών της. Απλώς σας εξηγούμε σε ποιο διαδικαστικό πλαίσιο λειτουργήσαμε. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1 του 2003, κάθε μέλος του δικτύου μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον θα ερευνηθεί μια υπόθεση ή όχι. Συνήθως ερευνάται ως προς την περίπτωση αυτή για την ελληνική αρχή ανταγωνισμού, τα αρχεία μας δείχνουν ότι αυτή έχει διεκπαιρεώσει πολλές υποθέσεις τα τελευταία χρόνια. 15 καινούριε μάλιστα που σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη δεν είναι λίγες. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί εδώ έχουν λυθεί από την ελληνική αρχή ανταγωνισμού εκτός από μία που η οποία βέβαια είναι σημαντική. Με συγχωρείτε κύριε μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν αλλάζει τίποτα από τη θέση μας. Θα γράψουμε λοιπόν επιστολή προς την κυρία Κρούς όπου θα τη ζητούμε να λάβει κάποια θέση. Ευχαριστώ τους αναφέροντες ή αναφερόμενους και ελπίζω να έχουν ικανοποιηθεί από την συνάντηση η κυρία Ματσούκα και ο κύριος Άτκινς έχουν δίκιο. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα γράψουμε επιστολή στην αρμόδια επίτροπο. Ε, λόγω πίεσης του χρόνου να πούμε ως Προεδρείο ε, ότι συμπαραστεκόμαστε στον απεργό πείνας, στον, για 77 ημέρες απεργό πείνας, κύριο Τενέζο, ε, και θα είμαστε δίπλα του στο δίκαιο αγώνα που καταβάλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατανοούμε το πρόβλημά σας, αλλά κλείνουμε εδώ αυτό το σημείο και πάμε, και πάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 18, λέει ο Πρόεδρος. Πέντε λεπτά έχει ο αναφέροντας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στερών. Και, ε, ποιο είναι το θέμα αυτό που μας απασχολεί. Είναι ε, εργοστάσιο εμφιάλωσης ε, μεταλλικού ύδατος στην Ισπανία. Έχουν παραβιάσει κάθε περιβαλλοντική νομοθεσία και σχετική νομοθεσία ισπανικές αρχές. Θα πρέπει να πούμε συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται. Δεν συμφωνούμε καθόλου με τα όσα ε, λέει η Επιτροπή σας και οι Ισπανικές Αρχές που λένε ότι μόλις το 0,2% ε, του υδροφόρου ορίζοντα είναι αυτό που θα εκμεταλλευτούν. Το ίδιο το εργοστάσιο μιλάει για 3,4 ε, κυβικά και εν πάση περιπτώσει αυτό που θα αντληθεί είναι το 45% του συνόλου και καθόλου αυτό που ορίζουν ε, ε, του ύδατος εκεί. Αυτό τι σημαίνει ότι το 1 τρίτο όρου του εμφιαλωμένου ε, νερού στην Ισπανία θα αντλείται από εκεί. Είναι πραγματικά εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Δεν συμφωνούμε καθόλου με την πρόταση αυτή ότι είναι μόλις το 0,2% Καθόλου. Είναι σχεδόν το μισό του νερού. 0,2% από όλη την υδρογραφική λεκάνη. αλλά όχι από το συγκεκριμένο ποτάμι. Και υπάρχει πρόβλημα φυσικά κατάντι. Έχουμε φέρει όλες ε, τις ε, απαραίτητες ε, δικαιολογητικές αναφορές και την οδηγία που αφορά τα ε, φυσικά μεταλλικά νερά. Δεν είναι όμως φυσικό μεταλλικό νερό γιατί έχει ε, υποστεί αφαλάτωση, ε, επεξεργασία με όζων και βακτηριολογική βελτίωση. Δηλαδή απάτη είναι τι μεταλλικό νερό προς τον καταναλωτή. Και υπάρχουν καταγγελίες προς τις ισπανικές αρχές οι οποίες υπεκφεύγουν και αποκρούν τις αναφορές μας. Και αυτό το συσκευαστήριο στον Τουρκάλ στην Ισπανία επίσης παραβιάζει τις οδηγίες για την περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την Άπιντατ και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Και πρέπει να σας πω ότι οι ίδιες οι αρχές γνωρίζουν και το αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται ε, μελέτη περιβαλλοντική παρόλο που δεν είχε γίνει ποτέ και ε, το αντίστοιχο ΙΓΜΕ της Ισπανίας, ε, το Μεταλλογικό Ινστιτούτο, θα αναγνωρίσει και αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ε, παραβίαση και στην πρόσβαση των αστικών υδάτων της κοινότητας και του Δήμου του Ντούρκαλ που θα αυξηθεί ο πληθυσμός του κατά 20% σύμφωνα με το αριθμιστικό σχέδιο και το πολυδημικό που ισχύει. Και με αυτά τα νερά και τόσα νερά που θα αντλούν για να τα αμφιαλώνουν, να τα κάνουν μεταλλικά, δεν πρόκειται να εξασφαλίζεται η υδροδότηση του πληθυσμού. Ούτε των εργοστασίων φυσικά που θα εγκατασταθούν εκεί. Και σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες επίσης ε, υπάρχουν ε, προβλήματα στα οποία θα αυξηθεί ο συνάδελφός μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι νοτίως της Γρανάδας, στο νότιο άκρο της Ευρώπης, έχουμε ε, μεγάλα προβλήματα με απειλούμενα είδη. Θα σας κάνουμε ακριβή έκθεση για να φορά και έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε και να καταλάβουμε ότι ε, θα πρέπει να μας υποστηρίξετε γιατί η Ισπανική κυβέρνηση ε, κοφεύει. Ευτυχώ που έχουμε, δόξα τω Θεού εδώ τον κύριο Χάμενστάιν και τον σύντροφο Βίλι Μάιερ. Θέλω να σα πω μόνο το εσεί. Ποτέ δεν πρέπει να λαμβάνετε καμία απόφαση για την κατανάλωση νερού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πλήρως οι επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει στο οικοσύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ pan Ο κύριος Χέλμουντ Μπλοχ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. If uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν μελέτησε πολύ προσεκτικά την αναφορά και τους νόμους, καθώς και τους ισχυρισμούς ότι ε, παραβιάζει την οδηγία για το, το για το νερό και την οδηγία για τα ε, οικοσυστήματα. Επίσης, την οδηγία για το εμφιαλωμένο νερό είναι μια οδηγία αγοράς, ε, δεν την ξέρω και θα πρέπει να επανέλθω. Για την προστασία της φύσης από τις πληροφορίες που έχουμε δεν προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για τα οικοσυστήματα, την οδηγία Habitat, γιατί δεν υπάρχει καμία απαγόρευση δραστηριότητας στην περιοχή και βλέπετε ότι ούτως ή άλλως ε, υπάρχουν οικοδομικές εργασίες όπως προβλέπει και οι τοπικές, προβλέπουν Για την οδηγία πλαίσιο για το νερό, το ποσό του νερού που χρησιμοποιείται ε, είναι αρκετά χαμηλό χαμηλή, μικρή ποσότητα. Επίσης υπάρχει, υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης ούτως ώστε να μην χαμηλώσει ο τροφόρος ορίζοντας λόγω της αφαίρεσης νερού. Αυτά τα δεδομένα τα έχουν όλοι οι πολίτες και με βάση την οδηγία για την πληροφορία για το περιβάλλον. Επίσης, ε, εξετάσαμε αν υπάρχει ε, παραβίαση ε, της οδηγίας για τη μελέτη επιπτώσεων. Όχι, γιατί η αφαίρεση νερού, το, το ποσό που αφαιρείται είναι πολύ μικρό. Επομένως, ούτε η οδηγία για τα οικοσυστήματα, ούτε η οδηγία για το πλαίσιο για το νερό, ούτε η οδηγία για την ε, μελέτη επιπτώσεων παραβιάζονται. Για την οδηγία για τα αφιελωμένα νερά θα επανέλθω με περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση της αυτή, διότι είναι γεγονός ότι από όλη την πληροφόρηση που μας έχουν δώσει οι ενοφερόμενοι, είναι υπάρχει κάτι που πρέπει να το λύσουμε. Τι εστί εφιαλωμένο νερό. Ε, ε, κανονικά πρέπει να είναι φυσικό μεταλλικό νερό, χωρίς καμία επεξεργασία. Απαγορεύεται κάθε είδους επεξεργασία. Αυτό το νερό εδώ τουλάχιστον τρεις επεξεργασίες έχει δεχθεί. Βακτηριολογική, με φίλτρα δηλαδή για τα μικρόβια, αφαλάτωση, ναι, απασβέστωση συγγνώμη, και το άλλο ε, οζόνωση Κανονικά λοιπόν είναι υποχρεωτικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει και να θεωρήσει ότι στρέφεται κατά του δικαίου του καταναλωτού. Θα πρέπει να μελετήσουμε εκτενέστερα και τις πληροφορίες αυτές για ενδεχόμενη χώριση του τμήματος Β ως μεταλλείο. Γιατί τότε είναι πραγματικά υποχρεωτικό να υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου για επιπτώσεων. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι έκτακτε οι περιστάσεις αυτού του εργοστασίου εμφιάλωση που είναι δίπλα στη Σιέρα ε, Νεβάδα που είναι ε, πραγματικά ένας τόπος που χρειάζεται προστασία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να μας ενημερώσουν και αυτή η ενημέρωση που μας δίνουν σήμερα αναφερόμενη να μελετηθεί με τον τρόπο που ζητούν εκείνοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάμερσεν Μίντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αγορά αλλά και η προστασία του καταναλωτού. Γι' αυτό θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αφορά και να το επιστήσουμε και την προσοχή της ισπανικής κυβέρνησης. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και στην επαρχία της Εγκόβια για παράδειγμα υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση. Δεπλόγια λέγεται το εργοστάσιο εκεί, νερό. Να ανοίξουμε, αφήσουμε ανοιχτή συγγνώμη αυτή την αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο εμπεριστατωμένη έκθεση. Μάλιστα. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό που είπαμε. Η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα περιμένουμε πρόσθετες πληροφορίες από την Κομισιόν. Ορίστε κύριοι αναφερόμενοι, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Δεν παίρνουμε την τελεϊκή μας θέση τώρα, όχι γιατί σας δίνουμε δίκαιο αναγκαστικά, αλλά γιατί δεν συμφωνούμε πλήρως με αυτά που είπε η Κομισιόν. Δεν συμφωνούμε δηλαδή ότι δεν υπήρξε παραβίαση των κανονισμών, των κανόνων. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, γι' αυτό παρακαλώ παραμείνετε σε επαφή και να μας πληροφορήσετε για τις εξελίξεις εάν υπάρξουν και θα μάθουμε και εμείς τι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το 14 όπου Έχουμε Βουλγάρους αναφερομένους από τον Εύξηνο Πόντο. Πρώτα η Κομισιόν και μετά οι αναφερόμενοι. Η κυρία Ποπόβα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι αναφερόμενοι με τις αιτήσει τους. Μερικές είναι από το 2007, άλλες από το 2008. Και από τότε έχουν σημειωθεί εξελίξεις στη Βουλγαρία ως προς τον καθορισμό των περιοχών Natura 2000. Σύμφωνα με τα, τις τελευταίες μας πληροφορίες η Βουλγαρία έχει καθορίσει 34% του εδάφους της ως, ως τέτοια περιοχή. Βέβαια χρειάζεται πολλά ακόμη να κάνει για την ταξινόμηση των κανόνων σύμφωνα με την οδηγία Brins. Έχουμε ταυτίσει έξι περιοχές για τα, για τα πετινά. Έχουμε καθορίσει έξι περιοχές και έγινε ένα σεμινάριο τον περασμένο Ιούνιο όπου ταυτίστηκαν ορισμένες ελλείψεις, όχι τεράστιες αλλά σημαντικές. Και από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 2009 πρέπει να μας δώσει όλες τις πληροφορίες η Βουλγαρία. Ούτως ή άλλως η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση και στάλθηκε και επίσημο γράμμα στην Βουλγαρία για την παραβίαση της οδηγίας των πετινών και Μόλις ετοιμαστούμε για την αξιολόγηση με βάση τις βουλγαρικές πληροφορίες θα δούμε τι μπορεί και πρέπει να γίνει. Το άλλο παράπονο των αναφερομένων είναι ότι αφορά μάλλον την ε, άδεια για ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Η Κομισιόν έμαθε από αναφορές ή από πρόσφυγες ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες επιτρεπόμενες δραστηριότητες στη Βουλγαρία και αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες αυτές. Μία από τις περιπτώσεις που είναι υποδειγματική θα έλεγα γιατί που δείχνει τι συμβαίνει στη Βουλγαρία είναι ότι η Κομισιόν διαπιστώνει Επανειλημμένος παραβιάσεις και έχουμε στείλει και γι' αυτό επιστολή. Για τις υπόλοιπες περιοχές ακόμη αξιολογούμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. Χρειάζονται και άλλα όμως για να δούμε κατά πόσον υπάρχει παραβίαση ή όχι. Και τέλος, έχω δει τις αναφορές, ιδίω για την Εμινέ, είναι η 1336 και είχαμε ζητήσει να παραταθεί η διορία εξέτασής της γιατί ακόμα περιμένουμε τις πληροφορίες. Είναι η μόνη αναφορά που δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε αλλά θα απαντήσουμε μόλις είναι έτοιμη, ίσως αρχές Ιουνίου. Σας κατευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε τέσσερις αναφερομένους εδώ στην αίθουσα. Κανονικά δίνουμε μόνο πέντε λεπτά στον καθένα. Αλλά ε, σε κάθε υπόθεση, αλλά πέντε λεπτά για τέσσερις είναι λίγα. Θα τους δώσουμε λίγο παραπάνω, αλλά παρακαλώ να είστε όσο δυνατόν συντομότεροι και συντομότερες. Η κυρία Βέρα Πετκάντσιν είναι εδώ. Πεντκάντσιν και μετά η κυρία Νέλια Αρμπατζίεβα. Με συγχωρείτε αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας, αλλά να τι να κάνω. Ο κύριος Κοβάτσεφ είναι και αυτός εδώ, ο κύριος Κοβάτσεφ. Σας οικετεύω να είστε συντομότατοι, ίσως ενάμιση με δύο λεπτά ο καθένας, γιατί πρόκειται για το ίδιο θέμα. Να μην ξεπεράσετε τα έξι λεπτά όλοι μαζί και όλες μαζί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κυρίες και κύριοι, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε διάφοροι αναφέροντες, γιατί το θέμα μας είναι κοινό. Ας ξεκινήσουμε την αφορά που αφορούν την ε, ακτή του εύξενου πόντου της ε, Βουλγαρίας και τις διάφορες παραβάσεις που γίνονται εκεί. Οι περισσότεροι από εσά θα γνωρίζετε την κατάσταση. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες εν εξελίξη σε διάφορα σημεία της Βουλγαρίας, δηλαδή ε, δασική γη ε, θεωρείται οικοδομήσιμη γη πια. Εξαιτίας αυτής της διαδικασίας λοιπόν και ενώ έχουμε αρκετά καλή κάλυψη από το Natura 2000 ε, στη Βουλγαρία. Στην πραγματικότητα δεν μας παρέχει προστασία ε, το Natura 2000 σε διάφορα σημεία της χώρας. Η παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα απλώς φύγει α, ακροφυγός τα πιο σημαντικά, τις πιο χοντρές παραβάσεις. Το 80% της ε, γης που καλύπτεται από το Natura 2000 είναι παράκτια περιοχή. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία από ένα φυσικό πάρκο στη Βουλγαρία. Υπάρχει μια, ε, ένας γενικός ε, χωροταξικός σχεδιασμός για όλη την ε, βουλγαρική επικράτεια. Όταν ο σχεδιασμός αυτός υιοθετήθηκε, δεν είχαμε λάβει υπόψη μας την επίπτωσή του στο περιβάλλον, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία της χώρας. Δυστυχώς αυτός ο σχεδιασμός είναι αναποτελεσματικός, ανεπαρκής. Αυτή είναι η μία από τις περιπτώσεις όπου έχουμε παραβιάσει από τη βουλγαρική κυβέρνηση. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία. Μία άλλη περίπτωση που έγινε πολύ γνωστή είναι η περίπτωση του Ιρακή. Εδώ βλέπετε την περιοχή. Σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Εδώ υπάρχουν οικοδομικές εργασίες. Σε αυτό εδώ το τοπίο. όλη αυτή η παραλία που βλέπετε θα χτιστεί. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ελπίζω ε, ότι θα μοιράσετε το χρόνο εργασίας μεταξύ σας. Έχω ακόμη τρεις ομιλητές. Δεν μπορείτε να μονοπολίσετε όλο το χρόνο ομιλίας. Κάποιος θα πρέπει να παραιτηθεί από το χρόνο ομιλίας του. Ναι. Ναι, ναι, θα συνοψίσω. Να πω δύο λόγια ακόμα για την περιοχή αυτή, το Ιρακή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν γίνεται σεβαστή. Ο κύριος Κοβάτσεβ. Ευχαριστώ. Θα, συζη... θα μιλήσω για αυτή την περιοχή, 5 χιλιόμετρα. Βρίσκεται δίπλα σε φυσικό πάρκο. Οι βουλγαρικές αρχές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καταστρέψουν αυτή την περιοχή φυσικής ομορφιάς και να την πουλήσουν σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν μάλιστα σε μια αυστριακή τράπεζα. Το 2007 η βουλγαρική κυβέρνηση επινόησε ένα πρόγραμμα για να χτίσει όλη αυτή την περιοχή και τα 5 ή 6 χιλιόμετρα παραλιακά χωρίς καμία αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και όλα αυτά έγιναν πολύ έτσι, ήσυχα ήσυχα, πολύ σιωπηλά, να μην το μάθει κανένας μέχρι να είναι πολύ αργά. Αυτό προσπάθησε να κάνει η βουλγαρική κυβέρνηση και το κατάφερε. Αύριο αυτή, αυτή η περιοχή, αυτό το πράσινο που βλέπετε, θα είναι καλυμμένο από τσιμέντο. Σε ό,τι αφορά το Καλιάκρε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Την έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της βουλγαρικής κυβέρνησης. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει συγκινηθεί και πολύ η βουλγαρική κυβέρνηση και γενικά οι βουλγαρικές αρχές δύο προγράμματα που είχαν εγκριθεί πριν ενταχθεί η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη δρομολογηθεί. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή οικοδομικές εργασίες. Ταυτόχρονα βεβαίως η, Ευρωπαϊκή, η βουλγαρική κυβέρνηση ε, ισχυρίζεται ότι προστατεύει τη φύση στη Βουλγαρία. Σας παρακαλώ, ο επόμενος ομιλητής, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν ακόμα 400 προγράμματα ε, τα οποία μπορούν να λάβουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν. Δεν πρέπει να περιμένουμε περισσότερο. Χρειαζόμαστε κατεπίγουσες ε, διαδικασίες όπως με τη Βία Μπάλτικα. Πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω για μια περιοχή ε, που προστατεύεται από το Natura 2000 στη Βουλγαρία. Ε, υπάρχουν εδώ φυσικά πάρκα. Βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Πρόκειται για την περιοχή της Ρίλα. Η Ρίλα, ενώ υποτίθεται εντάσσεται στο Natura 2000, ε, δεν προστατεύεται αρκετά. Υπάρχουν 8 ε, νέα ε, προγράμματα για χειροδρομικά κέντρα στο δρυμό της Ρίλα μέσα στον προστατευόμενο χώρο και γύρω από τον προστατευόμενο χώρο, σε αυτή την ουδέτερη υποτιθέμενη ζώνη. Αυτή η υποτιθέμενη ουδέτερη ζώνη στην πραγματικότητα είναι μία περιοχή που με βάση όλα τα επιστημονικά επιχειρήματα θα έπρεπε να είχε ενταχθεί στο Natura 2000 και να προστατευτεί απόλυτα. Δυστυχώς, χιλιάδες ε, προγράμματα και σχέδια έτσι, οικοδομικών κατασκευών και τα λοιπά έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ε, κοντά στη λίμνη, στις λίμνες της Ρίλα ε, πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες. Και μάλιστα και δίπλα σε ένα άλλο εθνικό πάρκο που είναι τμήμα του Natura 2000 θα γίνουν οικοδομικές εργασίες. Ε, αυτό το, πάρκο είναι ε, ενταγμένο και στις προστατευόμενες ζώνες της UNESCO. Εδώ υπάρχουν χιονονομικά κέντρα γύρω από τον Μπάνσκο και οι χιονοδρομικές ε, πίστες επεκτείνονται και μεγαλώνουν καθημερινά σχεδόν. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Βλέπετε την καταστροφή λόγω αυτών των κατασκευών, λόγω αυτών των οικονομικών εργασιών. Δεν υπάρχουν καθόλου μέτρα για να προστατεύσουμε τη διάβρωση του εδάφους, να προστατευτούμε από τη διάβρωση του εδάφους. Αυτά ήθελα να σας πω για αυτές τις υποθέσεις, για αυτές τις ε, περιπτώσεις και θα ήθελα τώρα να συνοψίσω. Ο τελευταίος ομιλητής, παρακαλώ. Ο πρόεδρος. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Η αναφορά μας αφορά και το δίκαιο ανταγωνισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Η βουλγαρική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκχωρεί δημόσια γη, την πουλάει, την απαλωτριώνει. Μιλάμε τώρα για δημόσια γη που βρίσκεται σε πολύ ελκυστικές περιοχές για τους επενδυτές και τους τουρίστες. Και η διαδικασία που υιοθέτησε η βουλγαρική κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα μια ανταλλαγή, ένας αποχαρακτηρισμός της γης. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την τοποθεσία αυτών των δημόσιων γεών. Σε ορισμένε περιπτώσεις ιδιωτικές γέες στην ενδοχώρα σε μη ελκυστικές τοποθεσίες για τους επενδυτές θεωρείται πολύ ακριβή, ενώ ταυτόχρονα η δημόσια γη σε παράκτιες περιοχές θεωρείται ως κάτι τρομερά φθηνό και μη ελκυστικό και το εκποιεί έτσι η κυβέρνηση. Δηλαδή, διαγράφονται πολύτιμα κομμάτια γης από το εθνικό κτηματολόγιο. Μιλάμε τώρα και για προστατευόμενες ακόμα περιοχές. Μερικές φορές η διαφορά στην τιμή μπορεί να είναι 280 φορές φθηνότερο ε, το κομμάτι της ε, δημόσιας γης. Δηλαδή η κυβέρνηση ξεπουλάει στην πραγματικότητα τη δημόσια γη και τη βγάζει στο σφυρί. Επομένως, οι απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Πρόεδρος. Κύριε Χριστόφ, θέλετε κι εσείς να μιλήσετε. Νομίζω δεν έχετε μιλήσει ακόμα, έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένας ακόμα ομιλητής. Ενάμιση λεπτό για τον τελευταίο ομιλητή παρακαλώ. Do you hear me? Yeah. Okay, thank you, Mr. Chairman, honorable members. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη. Θα τα πω αγγλικά μάλλον εγώ καλύτερα. Η βουλγαρική εταιρεία για την προστασία των πτηνών ε, και τη Ισπανίδα των πτηνών ε, έχει, ε, ακούσει, έχει πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει προσφυγή επί παραλήψη, αλλά δεν, κάνει, δεν θεωρεί επαρκή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ah, proszę bardzo, proszę kontynuować. Επανήλθε λοιπόν το σύστημα. Τώρα ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο κύριε Πρόεδρε. Δουλεύει. Καλούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λειτουργεί το μικρόφωνο του ομιλητού. Δεν λειτουργεί το φως, αλλά το μικρόφωνο δουλεύει. So, again, first accelerates infringement proceedings Bulgaria for failing to designate... Λέγω λοιπόν να ξεκινήσει αρχή ε, προσφυγή επί παραλήψης κατά της κυβέρνησης, αλλά κυβέρνηση αδρανή και θα πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες στη δικαιοσύνη για να σταματήσουν οι ζημίες που συνεχίζονται, για να σταματήσει ε, το συντομότερο η απώλεια της βιοποικιλότητας και να ξεκινήσει η προσφυγή στο δικαστήριο παραλήψη και να σταλούν και προειδοποιητικές ε, επιστολές για τη συνεχιζόμενη ε, ζημία τοποθεσιών που έχουν χαρακτηριστεί Natura 2000. Δεν υπάρχει επαρκή προστασία συστημική για τη Natura 2000 στη Βουλγαρία. Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη και πολλοί έκτακτες περιστάσεις και δεν μπορούν να ε, καθυστερούν οι διαδικασίες. Ευχαριστώ. Κυρία Στράφκοβα και μετά ο Χαμερστάιν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης καθώς και τη γραμματεία έχετε βοηθήσει πολύ τη Βουλγαρία να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και κατά τις επισκέψεις σας στη Βουλγαρία μας βοηθήσατε πολύ και ευχαριστώ επίσης τον Σερ Ρόμπερτ Άτκινς και τον κύριο Κόξ που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Για μένα θα ήταν εύκολο να σας πω ποια είναι η άποψή μου, αλλά και εσείς αφού πήγατε επί τόπου και είδατε τι γίνεται στη Βουλγαρία και στη βουλγαρική ύπεθρο και στη βουλγαρική φύση, τα ξέρετε. Υπάρχουν όμως μερικά καινούρια. Εγώ ζω στη Βάρνα που είναι λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα και δεν μπορώ να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια βλέποντας τι γίνεται εκεί. Με εκπλήσει ιδιαίτερα η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λένε ότι παρακολουθούν και θα αξιολογούν αυτά που γίνονται στη Βάρνα. Όσο παρακολουθούν όμως και όσο αξιολογούν καταστρέφεται η βουλγαρική φύση. Εμείς αναμένουμε από την Κομισιόν να ανταποκριθεί πιο συγκεκριμένα γιατί στην Σακτές της Βουλγαρίας συνεχίζονται οι καταστροφές. Οι ακτοί, ακόμη και τα βουνά καταστρέφονται και γι' αυτό σας ζητώ να λάβετε άμεσα μέτρα ώστε να δείξουμε ότι είμαστε στο πλευρό των πολιτών και όλων όσων ενδιαφέρονται για αυτά που γίνονται στη Βουλγαρία και ανησυχούν. Έχω εδώ στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία, τα γεγονότα είναι διαθέσιμα και σας παρακαλώ να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα, να ζητήσετε δηλαδή από την Κομισιόν να αλλάξει την αντιμετώπιση της. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια εκπρόσωπος της βουλγαρικής κυβέρνησης. Είχα ζητήσει να παραστεί κάποιος, αλλά δεν μπορούν γιατί υπάρχουν πολλές ε, αργίες αυτή την εποχή στη Βουλγαρία. Καλό θα ήταν να ακούσουμε τι έχουν και αυτοί να πούν. Ε, επειδή λοιπόν δεν είναι εδώ, εξαρτώμαστε από εσά, ο κύριος Χάμερστάιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας μιλήσω έξω από τα δόντια. Έξω. Σε ένα από τα ταξίδια μου στη Βουλγαρία, σε μια πρεσβεία μεγάλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάλεσε ε, ε όχι σε επίσημο εδαφός για να μου δει πώς αλλάζει η χρήση γης. Πώς αλλάζει η δημόσια γη ε, ε, και την πουλάνε χίλιες φορές περισσότερο και είναι Natura 2000. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τέτοια εκμετάλλευση. Είναι εκατοντάδες οι τόποι που προστατεύονται. Οι βουλγαρικές αρχές λένε ότι μπορούν να ε, μπουν στο σχέδιο ε, το πολεοδομικό οποιασδήποτε ε, περιφέρειες του, της φύσης 2000. Ας πούμε τα αγοράζει η γυναίκα του δημάρχου της Μόσχας σε υγροβιότοπους που είναι μοναδική χώρη αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αδρανεί με τρόπο σκανδαλώδη και απαράδεκτο. Και παρακαλώ τον πρόεδρο Λιμπίτσκι να πει ότι η Επιτροπή μας ζητάει διερεύνηση από πλευρά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού για την ολιγορία και απροθυμία για δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πιο μαζική καταστροφή. Εγώ Ισπανός είμαι και αισθάνομαι πάρα πολύ ε, ευαίσθητος γιατί αν ε, πριν από 20 χρόνια είχε αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχαμε ε, ε, τις ακτές που έχουμε σήμερα στην Ισπανία. Θα πρέπει να σώσουμε τον εύξηνο πόντο. Αν συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ω, μου το εξήγησε ο κύριος ε, Γκαρσία, ο αρμόδιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι μου λέει. Είναι εκατοντάδε οι παραβιάσεις μαζικές και κατάφορες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Α, οπότε διαλέξουμε μία. στη άκρα για να δράσουμε. Pick and choose. Όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά δεν έχει αυτή η υπόθεση το ε, χαρακτήρα διαπαιδαγώγησης που θέλαμε και παραδειγματισμού για να σταματήσουν τα υπόλοιπα έργα. Προφανέστατα δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι παραδειγματισμός αυτό. Πριν από δύο εβδομάδες πήγε όλα στη Βουλγαρία. Και μόλις κατέβηκαν από το αεροδρόμιο πιάσανε τους ταξιτζίδες για απάτη και τον ίδιο Υπουργό Μεταφορών ας πούμε. Καταλαβαίνετε η διαφθορά σε τι επίπεδα έχει φτάσει και η ασέβεια και η μη τήρηση των ε, συνθήκων των ευρωπαϊκών. Και είναι και παράδεκτη και απίστευτη η ολιγορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ χαίρομαι που η πολωνική κυβέρνηση ε, άλλαξε ε, τα δεδομένα της σύνθεξης βαλτικής, ε, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες ε, φορές χειρότερα είναι τόσο συμβαίνουν στον εύξηνο πόντο. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδρανεί, χίλιες φορές λιγότερο. Πώς αυτό εξηγείται. Εγώ θέλω να το ψάξει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Τι μεταχείριση επιφυλάσσουν στις καταγγελίες και στα γράμματα των οικολόγων της Βουλγαρίας και τι κάνουν με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, στρέφομαι προς την κυρία Στρακόφσκα και στον κύριο Χάμερστάιν Μίντς, που είναι και δύο ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να γράψουμε μία επιστολή προς την Επίτροπο Δήμα, έτσι μία πολύ αυστηρή επιστολή, και να τονίσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων στη Βουλγαρία. Ίσως καλύτερα να γράψουμε σε αυτόν παρά να γράψουμε στον διαμεσολαβητή. Καλύτερα να γράψουμε λοιπόν στον Επίτροπο. Δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει εμείς να απευθυνθούμε στο διαμεσολαβητή. Ίσως οι, οι ίδιοι αναφέροντες θα μπορούσαν να απευθυνθούν στο διαμεσολαβητή. Όχι, βλέπω τις χειρονομίες σας. Προτιμάτε να γράψουμε δύο επιστολές και στον Επίτροπο και στον Διαμεσολαβητή. Φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν οι αναφέροντες. Θα γράψουμε λοιπόν και στον κύριο Δήμα μία επιστολή και μία προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πάμε στο σημείο 21, 1448, κάθετος 2007. Ο κύριος Χένρικ Ντέμς, που είναι παρόν. Με μεγάλη χαρά σας βλέπω ήρθατε εδώ αυτοπροσώπως για να μας μιλήσετε για αυτό το ιστορικό μνημείο στην Πολωνία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους και τους διερμηνείς, λέει ο μιλητής. Αυτή η γέφυρα βρίσκεται σε μια δραματική κατάσταση. Ο Δήμος δεν έχει χρήματα και η κατάσταση χειροτερεύει ουσιαστικά από μέρα σε μέρα ζήτησε ακόμα και από την πολωνική κυβέρνηση να δώσει χρήματα. Με ένα εκατομμύριο θα σώζαμε τη γέφυρα. Η πολωνική κυβέρνηση μου είπε ότι πρέπει να παραιτηθώ από τις ελπίδες μου. Υπέβαλα και αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο. Διάβασα όλα τα έγγραφα τα οποία ετοιμάσατε. Το 2005 συντάχθηκαν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Τότε είχα επισημάνει το πρόβλημα στις αρχές. Οργανώθηκε μία διαβούλευση το 2007 για το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαζεμπόφσκι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος έστειλε ένα εμπειρογνώμονα για να διερευνήσει την υπόθεση και την κατάσταση από τεχνική απόψεως αυτή τη ιστορική γέφυρα στην Πολωνία. Θα ήθελα εσεί λοιπόν τώρα να ασκήσετε κάποια πίεση στις πολωνικές αρχές για να βρεθούν τέλο πάντων κάποια χρήματα. Είμαι θελοντής ε, και ασχολούμαι με την προστασία των ιστορικών μνημείων της Πολωνίας. Έχω γραφεί ακόμα και στο εξωτερικό και προσπαθώ εγώ ως εθελοντής να κάνω ό,τι μπορώ, ακόμα βγάζοντα και λεφτά από την τσέπη μου για να προστατευτούν τα εθνικά πολωνικά μνημεία. Πρόεδρος, καταλαβαίνω πόσο ανησυχείτε για την ε, κατάσταση αυτή τη ιστορική γέφυρα, αυτού του ιστορικού μνημείου. Εσεί μου τηλεφωνήσατε, πολλέ φορέ μάλιστα. Ε, μιλήσαμε για την κατάσταση της γέφυρας. Ε, εγώ είμαι πρόεδρος αυτής της επιτροπής, αλλά είμαι και ιστορικός τέχνης, ε, αυτό σπούδασα. Επομένως το θέμα αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που συζητούμε αυτό το θέμα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθώς και εμάς. Εμείς αναγνωρίζουμε όλα όσα έγιναν από τους εθελοντές για να σωθεί το μνημείο, αλλά η αρμοδιότητά μας για να παρέμβουμε σε αυτό το εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει. Το άρθρο 151 παράγραφος 2 είναι σαφέστατο ως προς τον περιορισμό των δικαιοδοσιών της Κομισιόν για την πολιτιστική κληρονομιά. Και η δικαιοδοσία δυστυχώς κύριε Ντέμς είναι, βρίσκεται στη συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών λέει οργανώσεων που λειτουργούν στην Ευρώπη. Όπως ίσως γνωρίζετε, στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά για να προωθήσει το θέμα. Και μία από τις δραστηριότητες της είναι και το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά, το οποίο πέρυσι έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε εκείνη τη γέφυρα στην Πολωνία. Και έγινε και μια ιδιαίτερη τελετούλα με εκείνη την ευκαιρία. Η ανταλλαγή λοιπόν πληροφοριών και τεχνογνωσίας είναι κάτι στο οποίο μπορεί να βοηθήσει η Κομισιόν, αλλά για χρηματοδότηση, για την αναπαλαίωση ή συντήρηση πολιτιστικών μνημείων τα κράτη-μέλη έχουν τη δικαιοδοσία. Ως προς την πολιτική συνοχή, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα μιλήσει γι' αυτό ο συνάδελφός μου, ο κύριος Πασούκ. Χαίρετε, θα μιλήσω παλαιονικά. Και εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία του μνημείου και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που κάνετε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εδώ που βασίζονται κυρίως στον κανόνα στην αρχή της επικουρικότητας. Εδώ το θέμα βρίσκεται στα χέρια των πολωνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρακολουθήσει παρά μόνο μεγάλου βεληνικούς ε, προγράμματα και όχι του μεγέθους που αφορά το δικό σας πρόβλημα. Κάτε μας, το πρόβλημα αφορά δύο προγράμματα. Πρώτο εκείνο που φέρει τον αύξοντα αριθμό 6 προτεραιότητος και υπάρχει εκεί μια θέση στον προϋπολογισμό για τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά όπου υπάρχουν 59 εκατομμύρια ευρώ και 44 είναι από την Ένωση. Στο εθνικό επίπεδο όμως θεωρητικά αυτό αφορά το πρόγραμμα υποδομές και περιβάλλον και υπάρχει προϋπολογισμός 560 εκατομμυρίων από τα οποία η Ευρώπη χρηματοδοτεί 490. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, ακούσαμε τα επιχειρήματά σας και καταλάβαμε ότι δεν είναι δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλα αυτά όμως, ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να σας πω ότι μας ανησυχεί η κατάσταση με την πολιτιστική κληρονομιά. Όποτε δηλαδή μνημεία καταστρέφονται ή βλάπτονται αυτό βλάπτει γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Γι' αυτό θα γράψουμε εν επιστολή προς τις πολωνικές αρχές όπου θα αναφέρουμε το πρόβλημα αυτό και τα επιχειρήματά σας και θα αναφέρουμε ότι μας ενδιαφέρει το θέμα και η γέφυρα αυτή και θα ζητήσουμε απάντηση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την απάντηση αυτή γιατί είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, το αυτό ήλπιζα κι εγώ. Μάλιστα, ωραία κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τον κόπο που κάνατε να προσέλθετε εδώ προσωπικά για να προστατεύσετε τη γέφυρα. Τώρα το σημείο 11. Αριθμός 471 κάθετος 2006 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπή. Για μια στιγμή. Έκανα λάθος. Το 12, το 12. 267-2007. Πρόκειται για σημαντικό στεγαστικό πρόγραμμα κοντά στο Ελσίνκι που κατά την αναφορά μπορεί να βλάψει το πρόγραμμα Natura 2000 μια περιοχή δηλαδή που έχει αναγνωριστεί εκεί κοντά στην περιοχή Κιβινόκα. Η αναφορά αυτή είχε ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή σας στις αρχές του 2007 και έγραψε επιστολή στις φιλανδικές αρχές που απάντησαν στις ερωτήσεις που είχατε θέσει και έδωσαν και περαιτέρω προφορίες για αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα. Η Κομισιόν αξιολόγησε το πρόγραμμα αυτό σε σύγκριση με το άρθρο 6 της Οδηγίας των Βιοτόπων και φάνηκε ότι το φινλανδικό σχέδιο πράγματι καλύπτει ένα τμήμα μιας περιοχής Natura 2000 και ότι μπορεί να βλάψει τον ε, πληθυσμό των πτηνών που κατοικούν εκεί. Επίσης λέει το πρόγραμμα ότι θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος εκεί και τον περιορισμό των ζημιών. Προβλέπονται αρκετά τέτοια μέτρα αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί από ό,τι γνωρίζουμε καμία απόφαση για την λήψη τους και προβλέπεται η περιοχή της Κιβινόκα την οποία για την οποία ενδιαφέρεται κυρίως η αναφορά θα συμπεριληφθεί στο φιλανδικό σχέδιο και πρόγραμμα και όλα αυτά θα εγκριθούν από την φιλανδική μεταφορά της οδηγίας των βιοτόπων. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει αυτό ή όχι και από ό,τι ξέρουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Φαντασόμαστε δε ότι οι αρμόδιες αρχές της Φιλανδίας θα εφαρμόσουν αυτά που μας δήλωσαν. Αν δεν το πράξουν βέβαια εμείς δεν θα ε, παραλείψουμε να κάνουμε προσφυγή. Χάμερστάιν. Παρακαλώ να διατηρηθεί η ανοιχτή αναφορά αυτή, είναι σημαντικό το θέμα. Υπάρχει και το προηγούμενο της υπόθεσης του Βοσαρή, θυμάστε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί αυτή η νομοθεσία, ιδιαίτερα για το οικιστικό ρυθμιστικό σχέδιο, διότι τραβάει σε μακρο αυτό και θα πρέπει να το προσέξουμε, να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Χάμερστάιν Μίντς. Πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά μετά από τις υποσχέσεις που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επανέλθουν περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε τον επόμενο μιλητή για το επόμενο σημείο τώρα, εδώ, που είναι το σημείο 13. Ε, έχουμε ε, ένα γύρι, γυριατρίο με 80 κρεβάτια ε, και την οικοδόμηση διαφόρων ε, κατοικιών ε, στην περιοχή μίας αλικής. Επίσης, η υπουργική απόφαση περιόριζε τον, την οικοδομική αυτή περιοχή. με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για τα ενδιατήματα. Αν υπάρξει επιρροή ε, αυτής της προστατευόμενης ε, περιοχής, ε, θα πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου να υπάρξει συντήρηση, διατήρηση αυτού του χώρου. Επίσης έχουμε και την οδηγία για τα πτηνά, την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε αν γίνεται σεβαστή. Έχει κοπεί το μικρόφωνο του ομιλητή. This one works. Θα αλλάξουμε θέσεις, γιατί το δικό μου μικρόφωνο δουλεύει. Τώρα με ακούτε, ωραία. Πολύ ωραία. Οι χώροι που προστατεύονται με βάση την οδηγία πτηνών θα πρέπει πριν από το χαρακτηρισμό τους ε, να ελέγχονται για να μην υπάρξει ε, επιδείνωση της κατάστασής τους και να μην διαταράσσεται ο χώρος που διαβιούν τα πτηνά. Η Κομισιόν έχει στείλει μία επιστολή στις Γαλλικές Αρχές τον ε, Ιούλιο του 2008 για να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει την αναφορά. Αυτές τις πληροφορίες, αυτές πληροφορίες όμως δεν έχουν ακόμα αποσταλεί στην Κομισιόν. Ε, στην ε, συνεδρίαση που κάναμε στο Παρίσι στις 6 Φεβρουαρίου του 2009 υπενθυμίσαμε αυτό το πρόβλημα. Η Επιτροπή σας θα ενημερώνεται από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λάβουμε τα έγγραφα από τις Γαλλικές Αρχές. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα να αφήσουμε και αυτή την αφορά ανοιχτή για να δούμε την προστασία ακριβώ των αλικών. Είναι ε, όλους διάζουσα αυτή η ακτή εκεί στην Κεράντ με τις αλικές. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα έτσι θα προχωρήσουμε και θα το διαβιβάσουμε στις αρμόδιες γαλλικές αρχές. αρχές. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο σημείο 15 κυρίε και κύριοι μου. 192 του 2006, κυρία Ισαμπέλ Λουρένκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για αυτή τον αυτοκινητόδρομο στην Ισπανία ε, δεν έχουν τελειώσει οι μελέτες περιβαλλοντολογικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Κομισιόν μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα λοιπόν δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστά. Και στις αρμόδιες ισπανικές αρχές πληροφόρηση για τα συμπεράσματα της μελέτης για να δούμε αν υπάρχει παραβίαση των περιοχών Natura 2000 και κατά πόσον η Ισπανία έλαβε υπόψη τις ε, τη ζημία που θα υποστούν οι περιοχές αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά κομμάτια. Περιμένουμε αρχές Ιουνίου την ισπανική απάντηση και όταν την έχουμε θα σας την υποβάλουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Χαμερστάν, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις απαντήσεις δεν μπαίνει στην ουσία της ερώτησης διότι η χάραξη και ο κορμός υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι η συνολική αξιολόγηση του ε, τμήματος, αλλά έχει κοπεί σε έξι κομμάτια και κάθε κομμάτι αφορά μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά είναι το ίδιο έργο στη χάραξη του. Και ο αντίκτυπος στα οικοσυστήματα είναι τεράστιος. Εδώ μιλάμε για τις εσχατιές της Ευρώπης. Είναι η ακτή απέναντι στο Μαρόκο, καταλάβατε την εκεί. Και είναι τα στενά του Γιβραλτάρ ε, με το φυσικό πάρκο εκεί. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Και το έχουν σαλαμοποιήσει για να κάνουν έξι διαφορετικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αυτό παραβιάζει κατάφορα την οδηγία. Επιπλέον, διότι δεν σταματάει εδώ, η έγκριση αυτή δόθηκε με διάφορα ονόματα. Η Α7 και η Α48 αυτοκινητόδρομος είναι ενιαίο πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι άλλο. Επιπλέον. Υπάρχει επέκταση αυτού του αυτοκινητοδρόμου, αλλά ορισμένα τμήματα του ήδη έχουν κατασκευαστεί και συνολικά έχουμε ε, πάρα πολλούς ε, βιοτόπους. Εκτελείται το έργο. Το έχω δει με τα μάτια μου τα ίδια τα έργα να γίνονται εκεί. Αυτή ο κατακαιρματισμός λοιπόν που το έχουν σπάσει για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη ε, τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στην οδηγία για τους οικοτόπους και τη σωρευτική του ε, δράση. Σκεφτείτε τα αυτά. Μιλάμε για πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Αν είχατε την τιμή να πάτε στην Ταρίφα στην Ισπανία ή στα στενά του Γιβραλτάρ. Είναι πολύ ιδιαίτερο το μέρος εκεί που ε, απειλείται και παρακαλώ να εφαρμοστούν ε, αμελητή και αυστηρά οι οδηγίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, θα πρότεινα λοιπόν να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά γιατί χρειαζόμαστε και περαιτέρω στοιχεία. Το επόμενο σημείο ο κύριος Χέλμουτ Μπλόχ θα μας ενημερώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω ότι πρόκειται για τον αριθμό 19, ε, ο κύριος ε, Τζόφρι Κέλτη Βρετανικής Ιδίας που δεν έχει σχέση με ε, τη μονάδα αυτή επεξεργασία των λιμάτων βιολογικού καθαρισμού πραγματικά ε, πρόκειται για παραβίαση της οδηγίας για τα αστικά λίματα και το βιολογικό καθαρισμό και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επί ε, παραδάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεταφορά της νομοθεσίας έχει γίνει σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει τελική ε, προειδοποίηση, αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης με δελτίο τύπου που να ενημερώνει τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης έχει ενημερώσει αρμοδίως και την Επιτροπή σας. Ωστόσο, ο αναφερόμενο επιμένει ότι αυτό είναι συγκάλυψη, συνωμοσία, συμπερνία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ισπανική κυβέρνηση ε, για να την απαλλάξουν από τις υποχρεώσεις τη. Αυτό αναφέρεται και σε μια πρόσφατη επιστολή προ εμάς κύριε Πρόεδρε που είχατε την καλοσύνη να τη διαβιβάσετε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να κατονίσει κανεί αυτέ τι αιτιάσει. Έχουμε ξεκινήσει την ένδικη διαδικασία και απειλούμε το κράτος μέλος ότι θα πάμε στα δικαστήρια. Αυτό είναι συγκάλυψη ή ναι. συνωμοσία για να την απαλλάξουμε των ευθυνών της. Μάλλον το αντίθετο είναι. Συνοψίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για την πληροφόρηση ε, που απορρέει από την Επιτροπή σας και έχει αναλάβει νομικά. Στο παρόν έχουμε ακριβώς την ε, αιτιολογημένη γνώμη και θα ακολουθήσει και το δικαστήριο. Όχι μόνο για το Λομπριγκάτο αλλά και για άλλα άλλους δήμους και κοινότητες αν χρειαστεί. Εξετάζουμε τα επόμενα βήματα και μπορεί να φτάσουμε και μέχρι το 10. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δίνει συνέχεια. Ελπίζω να αυτό φτάσει και μέχρι το 10. Προφανώς το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ερχόμαστε εκ των υστέρων για να ε, κάνουμε την νεκροψία. Η συγκεκριμένη ε, αναφορά είναι από το 2006. Έχουν περάσει από τότε πάνω από τρία χρόνια. Και η συγκεκριμένη περίπτωση ε, που μας απασχολεί συνεχίζεται. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ σωστά αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δραστήρια και εφαρμόζοντα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, πάμε στο επόμενο σημείο, 20. Και πάλι ο κύριο Βλόχ. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή αφορά τη μόλυνση του ποταμού Χούκα στην Ισπανία. Είναι γνωστός ποταμός για τους περιβαλλοντολόγους καθώς και τους γεωργούς και τους δήμους. Έχει πολύ υποφέρει. Έχουν υποφέρει και τα ψάρια. Και όπως λένε και στην αναφορά, η μόλυνση αυτή οφείλεται στο ότι στον ποταμό αυτό χύνονται ακάθαρτα ύδατα ή μη καθαρισμένα ύδατα. Γι' αυτό η Κομισιόν προσέφυγε. Ανάλογα και με την περίπτωση της Κορδέρα του Λιουμπρεγκάτ. Έκανε την τελική δηλαδή προειδοποίηση πριν από προσφυγή στα δικαστήρια. Αν δεν διορθωθεί η κατάσταση τους επόμενους μήνες θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Πράγματι, αυτός ο ποταμός Χόκαρ ε, ρηπαίνεται πάρα πολύ. Ρήπανση. Ε, στο δεύτερο μεγαλύτερο υγροβιοτοπό, ένα φυσικό πάρκο της Λαβουθέρα, μια σειρά δήμων και κοινοτήτων άνω των 10.000 κατοίκων δεν διαθέτουν ε, ε, διολογικό καθαρισμό των λιμάτων και θα γίνουν στο ποτάμι. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κοιτάζει και το αντιμετωπίζει οριζόντια, αλλά πολλές φορές αυτές οι οριζόντιες διαδικασίες δεν είναι αποτελεσματικές και χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Στην περιοχή εκείνη έχουμε ήδη ε, απόφαση του ΔΕΚ για τα απόβλητα στην Μωτίγια ε, και Σουέκα που είναι παραλίες δίπλα και βλέπουμε να ψοφάνε τα ζώα, να πεθαίνουν τα, τα, τα ψάρια. Είναι Natura 2000 φυσικών πάρκων και ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Ε. Έτσι. Και παρόλα αυτά ο δήμαρχος αυτού του χωριού που λέγεται Σουέκα, ότι αφού δεν μας βάλανε πρόστιμο ε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνω βιολογικό καθαρισμό. Αυτό το λέει ανοιχτά στον τύπο. Εγώ ενημέρωσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επιθυμούσα ε, προφανώς να ξαναπευθυνθείτε στο δικαστήριο για την παραλία αυτή στη Μωτήγια που είναι το ίδιο ποτάμι και να επιληφθείτε του θέματος γιατί από ό,τι φαίνεται ο Δήμαρχος κοφεύει. 40.000 30-40 και κάτοικοι, δεν έχουν λεφτά για να βάλουν βιολογικό καθαρισμό. Λέει αφού είναι δωρεάν, αφού δεν έχει πέσει κανένα πρόστιμο, δεν πειράζει, ας το έτσι. Παρόλο που υπάρχει σαφέστατη καταδικαστική απόφαση. Ευχαριστώ. Και προχωρούμε. 22. Ο κύριος Μιχαήλ Μεντούνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την αναφορά αυτή την ανέλαβε ο πρώην συνάδελφός σας Λόρδος Ίγκολγουντ που μίλησε για άνηση μεταχείριση και είπε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα της διπλής απασχόλησης των Λόρδων ως Ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με ένα νομοθέτημα του 76 για τις εκλογέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η θέση, ή μάλλον η θέση ενός εθνικού βουλευτού θεωρείται πλέον ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού. Και γι' αυτό πρέπει και στο Ηνωμένο Βασίλειο να λυθεί το πρόβλημα αυτό πριν τις ευρωεκλογέ. Η κυβέρνηση προσπάθησε να εισαγάγει αυτό το νέο νομοθέτημα για τη Βουλή των Λόρδων, αλλά έτσι έδωσε τη δυνατότητα σε έναν ισόβιο Λόρδο να παρετείται από τη Βουλή των Λόρδων κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τους κληρονομικούς Λόρδους. Γιατί στη Βουλή των Λόρδων υπάρχει ένας εγγυημένος αριθμός κληρονομικών Λόρδων κατάλογος που έχει ταρτιστεί από το 92 τουλάχιστον και θεωρείται ότι υπάρχει άνηση μεταχείριση λοιπόν μεταξύ των δύο ειδών λόρδων ισοβίου και κληρονομικού. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η Κομισιόν έλαβε, έχει πολύ λίγο χρόνο που έλαβε την αναφορά αυτή και δεν μπόρεσε να κάνει μια επίσημη γνωμοδότηση. Αυτά που σας λέω εδώ είναι προκαταρκτικά. Κατά πρώτον φαίνεται ότι πράγματι η μεταφορά του νόμου αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο που δίνει τη δυνατότητα στους ισόβιους λόρδους να παρετούνται αλλά όχι για τους κληρονομικούς είναι πράγματι αντίθετη με τον νόμο του 76 και η Κομισιόν σχεδιάζει να έρθει σε επαφή με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να διασφαλιστεί ότι προσεχώς στις ευρωεκλογέ δηλαδή, στις προσεχείς ευρωεκλογέ θα λυθεί αυτή η διαφορά μεταξύ ισοβίων και κληρονομικών λόριδων. Θα ήθελα να ζητήσω από τον David Law να μας μιλήσει, γιατί μίλησε με Inglewood. Θα ήθελα να σας πω σε όλους τους συναδέλφους που είναι παρόντες εδώ ότι επειδή ο Λόρδος Ίγκολγου δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, μου έδωσε, μου έστειλε ορισμένα έγγραφα και ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε που αναλάβατε τόσο σοβαρά το θέμα αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής μας έλαβαν το αντίτυπο μιας νομικής γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου και το πρωί και την επίσημη γνωμοδότηση της Επιτρο... Θεσμικής Επιτροπής που είχε εξετάσει επίσης αυτό το θέμα και τα συμπεράσματά τους νομίζω συμφωνούν με την πρώτη μας συζήτηση να γράψουμε δηλαδή στον πρόεδρο της Βουλής των Λόρδων που είναι και μέλος της κυβέρνησης για να τονίσουμε την ύπαρξη του προβλήματος και να ζητήσουμε εξηγήσει για το πώς εξηγείται αυτή η διαφορετική μεταχείριση των δύο ειδών λόρδου. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο το 23. 567 κάθετος 2008, ο κύριος Γαβριάδης. Ευχαριστώ. Η αναφορά αφορά την άρνηση του φλαμαδικού κέντρου, ακτινολογικού κέντρου να δώσει αντίτυπο στα γαλλικά. Ε, για τις δύο ακτολογικές εξετάσεις που έκανε ο αναφέροντας. Ε, ο αναφέροντας αναφέρει ότι μια και το Βέλγιο είναι μια τρίγλωση ε, γλώσσα, χώρα, θα πρέπει κανονικά να δίδονται τα έγγραφα και στα γαλλικά. Η απάντηση της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη. τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των γλωσσών, τη χρήση των επισήμων γλωσσών στο Βέλγιο καλύπτονται αποκλειστικά από την εσωτερική ε, συνταγματική τάξη του Βελγίου και δεν έχουμε τίποτα περαιτέρω να προσθέσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ε, σαφής η περίπτωση και μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή. 24 του 2002, ο κύριος Δανιέλ Βάρα έχει το λόγο.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 Proszę Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο ε, αναφορών στο σημείο Α και όχι μόνο. Τώρα έχουμε όμως αναφορέ στο σημείο Β ε, και κλεισμένων το θυρών όμως. Με εξαίρεση εκείνους που Έλαβα διαφορετική απόφαση. Προτείνω λοιπόν τώρα να περάσουμε στα σημεία Β, αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φόντ της γραπτής απάντησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επόμενη όμως αναφορά πρέπει να πάει στο Α, όχι το Β. να σταματήσει εδώ η συνεδρίαση σήμερα, να την κλείσουμε. Ευχαριστώ όλους τους ε, συμμετέχοντες της εργασίες και με μεγάλη ικανοποίηση είμαι σε θέση να σας πω ότι ο David Hammerstein Mintz είναι ο επιμελέστερος και από τα δραστηριότερα μέλη της, Επιτροπής μας και τώρα που ολοκληρώνονται οι ε, συνεδριάσεις μας. Ποιος έχει απομείνει, ο κύριος Χάμερστάιν Μίντς. Σας ευχαριστώ όλους και ε, ιδιαίτερο στη γραμματεία και δεν μπορώ παρά να τονίσω κάτι που έχω ξαναπεί. Η γραμματεία ήταν πάντα υπερκομματική και αν με ρωτούσε κανείς τι πολιτικών πεπιθήσεων είναι ο Ντέβιτ Λόου, έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Διότι η γραμματεία πραγματικά ε, δούλευσε πάντα επί της ουσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς όλους τους εκπροσώπους της που συμμετείχαν με πάρα πολύ δραστήριο και ενεργό τρόπο στις εργασίες της Επιτροπής μας πάνω από πέντε χρόνια. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες μας τώρα δεν θα μπορούσαμε να ε, δουλεύουμε χωρίς τη γνωμοδότησή σας, αλλά θέλω να πει κάτι ο κύριος Χάμερσταϊν Μίντς. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε ο οποίος ήσασταν και γενναίος και αμερόληπτος και στεναρός πρόεδρος. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει, ε, να έχουμε διεκπαιρεώσει τόσο μεγάλο ρυθμό αναφορών. Και βεβαίως πρέπει να συγχαρώ και τη γραμματεία, η οποία δούλεψε πραγματικά έντονα σε δύσκολες συνθήκες, ε, ανεπαρκώς τελεχωμένη, με κατακλυσμένη από πληθώρα αναφορών, με πολλές επικρίσεις από δεξιά και αριστερά. Θέλω να συγχαρώ και άλλους. Είμαι ο μόνος ευρωβουλευτής, αλλά δεν πειράζει, γιατί υπάρχουν εδώ και κάποιοι αναφέροντες. Θα ήθελα να τους ε, ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έμειναν εδώ και που το δείγμα τους είναι αντιπροσωπευτικό και συμβολίζει τους ανθρώπους, το καλύτερο τμήμα από αυτούς που πέρασαν από αυτή την Επιτροπή. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν βάλει και με γίγαντες, δεν, φοβούνται κανένα. Αυτή ήταν η στάση όλων μας, ε, η στάση σας πρόεδρε και η στάση της γραμματείας. Πρόκειται για δημοσίους, δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν το, τη δουλειά τους σαν ένα λειτουργήμα και δεν είναι σε διακοπές. Πρόεδρος, θα ήθελα να τα καταγράψουμε όλα αυτά στα πρακτικά και τις, ε, τα καλά σας λόγια και τα κοπλιμέντα. Τίποτα να μην λείψει. Σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να κλείσω αυτό το, αυτή τη συνάντηση. Άλλο ο Πρόεδρος ευχαριστεί πολύ γενικά και τους διορμηνείς. Και εμείς βεβαίως.